Uh, λοιπόν, καλησπέρα σας. Συγγνώμη που καθυστέρησα κάπως. Ασυνήθιστο. Αλλά είχε μια τεράστια, είχα μια τεράστια ομάδα που να με δει και καθυστέρησα. Λοιπόν, έγκριση μεσίας διάταξη. Δεν διαφωνεί κανένα. Και ήθελα να κάνω μια μικρή αλλαγή τι ανακοινώσει του Προέδρου Λετερίνα τι κάνουμε αργότερα για να περάσουμε αμέσως στην ανταλλαγή απόψεων με τον Τζόρι Ακερχόλμ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για την Διακυβέρνηση των τομέα της στατιστικής. Τη ΕΦΚΑ, που από ό,τι θυμάμαι γι' αυτό το σώμα ήμουνα κάποτε στην περασμένη δεκαετία εισηγήτρια. Πόσο θα σας δώσουμε, 10 λεπτά για την εισαγωγική σας ε, παρατήρηση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ γενναιόδοροι είσαστε. Α, πέντε λεπτά λέει η Πρόεδρος. Να δούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η τρίτη και τελευταία έκθεση για το SK1. Η εντολή μα ε, λύγει τον επόμενο μήνα και έχει οριστεί μια νέα επιτροπή και γι' αυτό ήθελα να σχολιάσω την γενική εμπειρία μας και να μπούμε μετά στις λεπτομέρειες της έκθεσης που έχει υποβληθεί. Σε γενικές γραμμές έχουμε την εντύπωση ότι έχει σταματήσει η πρόοδος υπήρχε κάποια πρόοδος από τότε που σας παρουσίασα τα πράγματα πριν από ένα χρόνο, αλλά πολλά ακόμα μπορούν να βελτιωθούν. Συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας σε τρεις αρχές. Επαγγελματική ανεξαρτησία, διαθεσιμότητα πόρων και ποιότητα. Άμα τα σκεφτείτε, θα δείτε ότι είναι πολύ σημαντική για το βάσιμο των στοιχείων αλλά επίση δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι τα πρώτα δύο, δηλαδή η πόρη και η επαγγελματική ανεξαρτησία, δεν είναι στα χέρια των στατιστικών υπηρεσιών. Είναι κάτι που αποφασίζεται σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό που κάναμε είναι ότι μια που έχουμε περιορισμένους πόρους, ε, χρειάστηκε να συγκεντρωθούμε και να μπούμε περισσότερο εις βάθος στα θέματα που θεωρούμε σημαντικά. Η πρώτη μας έκθεση βασίζεται στις πληροφορίες που μου δίνει η Eurostat. Δεν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε πολλά άλλα πράγματα. Μέχρι τότε η δεύτερη έκθεση βασίστηκε σε αυτά συν το ερωτηματολόγιο προς τα εθνικά στατιστικά Ινστιτούτα και κάποιους από τους άμεσα Κάτι που μας έδωσε πιο ευρία βάση για αξιολόγηση. Συνεχίσαμε στην ίδια βάση και για την τρίτη έκθεση, αλλά είχαμε ένα διάλογο για 8, ε, με οκτώ χώρες και με τα Ινστιτούτα ΕΣΚΑ Μπλοκ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία. Το πιο δυσάρεστο ήταν ότι μάθαμε ότι δεν είναι το ίδιο η πράξη και η θεωρία. Ό,τι υπάρχει σε χαρτί είναι ένα πράγμα. Απ' την άλλη μεριά, στην πράξη παρουσιάζονται πολλά προβλήματα. Ε, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση της διακυβέρνησης, δηλαδή αναθεώρηση του κώδικα συμπεριφοράς και χαιρετίζουμε επίσης τα στοιχεία στην ανακοίνωση για πιο ισχυρή διαχείριση της πολιτικής και επίσης χαιρετίζουμε τις προσπάθειες ούτως ώστε να τμήμα του κώδικα να περάσει στην νομοθεσία. Πράγμα που δίνει περισσότερη ισχύ στην Κομισιόν. το 60% των μέτρων που είχαν ε, σημειωθεί στην peer review αυτή, στην εξολόγηση ισοτήμων, έχουν εφαρμοστεί. Ορισμένες χώρες ε, δεν έχουν δώσει τα στοιχεία, ε, άλλες συνεχίζουν τώρα να εξυγχρονίζουν. και μια, υπάρχει και μια βελτίωση στον καθορισμό των παρατορεοτήτων. πολύ σημαντικό γιατί δεν έχουμε και τόσο πολλούς πόρους. Όσον αφορά την ποιότητα υπήρξε κάποια πρόοδος, να πούμε και κάτι θετικό για την Ελλάδα. Υπήρξε ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ελστατ και άλλων ε, υπηρεσιών στατιστικών στοιχείων. Στη Σουηδία υπάρχει τώρα ένα σύστημα ε, προπονητών, αν θέλετε, ποιότητας, quality coaches, Επίσης είδαμε ότι υπάρχει καλύτερη συνεργασία με τη Βουλγαρία και με την Τσεχική Δημοκρατία. Τούτου λεχθέντος όμως, μετά από πέντε χρόνια εφαρμογής, το 40% των μέτρων δεν έχει εφαρμοστεί. 275 ε, μέτρα συγκεκριμένα δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα και αν δεν είναι όλα ίσης σημασία, παρόλα αυτά είναι ε, αυτή η κατάσταση και πιστεύουμε ότι χρειάζεται περισσότερη πολιτική προσπάθεια για να προχωρήσουμε. Όσον αφορά την επαγγελματική ανεξαρτησία, σημειώσαμε ότι υπάρχουν ορισμένες χώρες, μεταξύ αυτών και η Δανία, όπου η πρακτική ίσως είναι σύμφωνη με τον κώδικα, αλλά όχι η νομοθεσία. Και θα πρέπει να προσαρμοστεί η νομοθεσία, κάτι για το οποίο δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχέδια. Λυπηρό. Επίσης, στη Σουηδία βλέπουμε ότι σε ορισμένες χώρες όπως στη ε, Λετωνία, Γερμανία, Ελλάδα, η εφαρμογή δεν προχωρά όπως θα έπρεπε. Και μάλιστα ε, πρόεδρος έστειλε μια επιστολή στην Ελλάδα που φαίνεται ότι κάπου χάθηκε όμως γιατί δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση. That uh, Λυπούμεθα ότι δεν είναι διαφανής η μέθοδη πρόσληψης και απόλυσης στις εθνικές ε, στατιστικές υπηρεσίες υπάρχει ένα πρόβλημα με διαδικασία στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Δεν κατηγορούμε κανένα βέβαια. Από την άλλη μεριά θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείται οπωσδήποτε η εμπειρία. Πόροι. Αυξάνουν τα προβλήματα. Για λόγους ευνόητους. Δεν νομίζουμε ότι είναι πολλά υποσχόμενο να ζητήσουμε περισσότερους πόρους για τις στατιστικές υπηρεσίες. Εμείς προσπαθήσαμε να υποβάλουμε κάποιες ιδέες για να γίνουν εξοικονομήσεις στη χρήση των πόρων. Αυτά τα μέτρα προβλέπουν ε, πιο έντονη συνεργασία πέρα από τα εθνικά σύνορα. Και θα θέλαμε επίσης να υπάρχει ορισμός ερωτήτων. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να δούμε επίσης τις επενδύσεις. Γιατί πολιτικά είναι εύκολο ε, να πα... Ε, γίνουν περικοπές στις επενδύσεις και όχι στις τρέχουσες ε, δαπάνες. Προσπαθήσαμε να ενώσουμε τις επενδύσεις σε τρεις ομάδες, γνωρίζοντας ότι κανένας δεν επιτρέπεται να περικόψει τις επενδύσεις που έχουν σαν στόχο ου εκείνε που έχουν σαν στόχο την βελτίωση της ποιότητα, αλλά εκεί που έχουμε νέου τομείς πρέπει να είναι κανένα προσεκτικό. Προτείνουμε επίση ότι θα ήταν ίσω χρήσιμο να εισαχθεί προπολογισμό πολυετή στον τομέα αυτό για να είμαστε σίγουροι ότι δεν απειλούνται οι επενδύσεις. Για την Ευρωστάτ ε, προτείνουμε τον εξορισμό της απόφασης της Κομισιόν του 1997 που ορίζει το ρόλο της Ευρωστάτ και ενθαρρύνουμε την παρακολούθηση των πρωτοβουλειών που έχουν σαν στόχο την ενδυνάμωση των ε, κρατικών δομών. Επίσης αναμένουμε ότι οι προβλεπόμενες αλλαγές στην εσωτερική οργάνωση της Ευρωστάτ που θα μειώσει το προσωπικό από 50 σε 45 και θα αυξήσει τους ελέγχους που γίνονται στους τομείς της διαδικασίας έλλειψης. Πολύ χρήσιμο. Κυρία Πρόεδρε, δύο λόγια για το τι μάθαμε από τα πρώτα αυτά χρόνια της λειτουργίας του ΕΣΚΑΠ 1. Το πιο σημαντικό είναι ότι είχαμε την εντύπωση ότι υπήρχε ένα κενό μεταξύ των προσδοκιών για την ΕΣΚΑΠ και αυτών που είδαμε ότι θα μπορέσουμε να προσφέρουμε τελικά. Και αυτό που αποφασίσαμε είναι να προσαρμόσουμε τα αποτελέσματά μας στους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Και έτσι να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στα πιο χρήσιμα αλλά ομολογώ ότι εγώ θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να υπάρχουν κάποιες διευκρινήσεις για τις ε, προσδοκίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τα αποτελέσματα της εργασίας της ΕΣΚΑΠ. Γιατί είναι καλό να λέμε ότι έχουμε ένα κώδικα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι η ΕΣΚΑΠ. Αλλά όταν πούμε ότι έχουμε έναν κώδικα και έχουμε και την ΕΣΚΑΠ η οποία φροντίζει να εφαρμοστεί 100% ο κώδικα αυτός, βρισκόμαστε σε κάποιε δυσκολίε. Γιατί δεν θα πούμε την αλήθεια αν πούμε ότι έχουμε ένα σύστημα το οποίο προσφέρει αυτά που θέλουμε. Η ΕΣΚΑΠ έχει 7 μέλη, επαγγελματικά μέλη που δεν πληρώνονται και ένα μέλος γραμματείας. Αυτό βέβαια περιορίζει τις εργασίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ε, μια βάση πληροφοριών, αλλά μάθαμε επίσης ότι για να μπορούμε να είναι πραγματικά αποτελεσματικοί, πρέπει να μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα. Πρέπει δηλαδή να μπορούμε να κατονομάσουμε τα προβλήματα που βλέπουμε. Ε, καταρχήν αποφασίσαμε να μην κατονομάζουμε χώρες. Γιατί πιστεύουμε ότι δεν είχαμε τις ε, βάσεις πληροφοριών να το κάνουμε αυτό. Τώρα πια όμως μπορούμε να κατονομάσουμε χώρες όταν πρόκειται για συγκεκριμένα στοιχεία και υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις όχι πολύ αλλά κάποιοι τέλο πάντων. Ιδανικά βέβαια θα πρέπει κάποιος να μπορεί να κατονομάσει κάποιο πρόβλημα που θεωρεί ότι υπάρχει, που δεν βασίζεται σε δεδομένα, αλλά σε κάποια γνώμη, σε κάποια ιδέα. Αυτό προβλέπει όμως πολύ πιο βάσιμη βάση πληροφοριών από εκείνη που μπορεί να δώσει η ΕΣΚΑ αυτή τη στιγμή. Και θα πρέπει βέβαια να φροντίσουμε να μην γίνει κανέναν λάθος στη διαδικασία αυτή. Κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ίσως υπάρχουν διαφορά μεταξύ θεωρίας και πράξης και ότι χρειάζονται πάρα πολλέ πληροφορίε για να μπορεί κανένας να κρίνει τι γίνεται στην πράξη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κάποιος να μπορεί να εμβαθύνει πάρα πολύ για να μπορέσει να δώσει μια καλή βάση πληροφοριών για να μπορεί να κάνει τις σωστές ε, εκτιμήσεις αλλά κάναμε ό,τι μπορούσαμε και προσαρμοστήκαμε σε αυτό που είχαμε στα χέρια μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Σοφή. Θέλεις να πάρεις το λόγο. Υπάρχει κανείς άλλος. Ο κύριος Χοντής, άλλος. And, and, and Okay, so I'll, well, I'll take you in the order which indicated. Θα πάρετε το λόγο με τη σειρά που σημειώσαμε. Σοφή, παρακαλώ. Yes, thank you, Madam Chair. Maybe the rapporteur wants to come in. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μήπως ο εισηγητής θέλει πρώτος να παρέμβει. Όχι. Ε, σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ε, αποκτώ την εντύπωση ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δύο σύντομες ερωτήσεις έχω, τρεις. Η πρώτη είναι... Συνδέεται μάλλον με το, το, το σύστημα θα πρέπει να οριμάσει και να αναπτυχθεί. Είσαστε αισιόδοξο ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί σύντομα. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με τη Eurostat. θα λέγατε ότι ακόμα με τις αλλαγές που αναφέρατε η Eurostat ε, θα πληρεί τα δικά σας πρότυπα ανεξαρτησίας. Ή πιστεύετε ότι θα είναι απαραίτητη μια αλλαγή του νομικού καθεστώτος ή του θεσμικού καθεστώτος της. Ε, και η τρίτη μου ερώτηση όσον αφορά τα δημοσιονομικά. Πώς βλέπετε την συνεργασία με ε, τα Εθνικά και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω τώρα που θυμάμαι ακόμα την ερώτηση. Είμαι αισιόδοξο. Ε, θα είμαι αισιόδοξο εφόσον υπάρχει περισσότερη ε, ε, πολιτική υποστήριξη. Χρειάζεται μια όθηση για να ανακτήσουμε την ταχύτητα που είχαμε αρχικά το 2005-2006 ίσως και το 2007. Όταν κάναμε εμείς αυτή τη δουλειά, νιώσαμε ότι οι εργασίες αυτές δεν έχουν λάβει την προσοχή που έπρεπε να έχουν λάβει σε εποχή κρίσης και όλας. Καταλαβαίνω γιατί έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να θυμόμαστε όμως ότι οι στατιστικές μας έχουν δημιουργήσει και όλας πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο θέλουμε να λύσουμε, να μην δημιουργήσουμε νέα προβλήματα. Χαίρομαι με τις αλλαγές που έχουν γίνει και αυτές που γίνονται και που σχετίζονται με τη Eurostat. Θεωρώ χρήσιμο να δούμε πώς θα λειτουργήσουν τα πράγματα αυτά, προτού να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε νέες αλλαγές. διότι νομικά μπορούμε να υποφεληθούμε και από το γεγονός ότι η Eurostat αποτελεί μέρος της Κομισιόν. Αυτό της δίνει κάποιες εξουσίες. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Όσον αφορά τη συνεργασία με τους ελεγκτές, υπάρχουν κάποια υπέρ και κάποια κατά. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Φυσικά υπάρχουν δυνατότητες εξορθολογισμού όσον αφορά την πληροφοριακή βάση. Θα πρέπει όμως να θυμόμαστε επίσης ότι οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς στόχους και δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε την ε, κατάσταση όπου στατιστικές ε, χρησιμοποιούνται για νομικούς στόχους ε, ή για στόχους ελέγχου, διότι αυτό θα δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων και την ευθύνη στην περίπτωση αυτή. Θα πρέπει να γνωρίζουμε δηλαδή τους πιθανούς κινδύνους. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε εισηγητή για το θέμα αυτό. Πρόκειται απλά για ανταλλαγή απόψεων. Και γι' αυτό χρησιμοποιούμε το σύστημα Catch the Eye. Ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Άκερχολμ για την ενδιαφέρουσα ε, παρουσίαση που μας έκανε κατάλαβα ότι έχει μια συμπυκνωμένη εμπειρία για τα ευρωπαϊκά στατιστικά. Γι' αυτό θα ήθελα να το ρωτήσω τα εξής πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, είμαι από την Ελλάδα και αναφερθήκατε ορισμένες φορές στην εισήγησή σας κυρίως ότι ακόμα οι ελληνικές αρχές δεν κάνουν αυτά που θα έπρεπε να κάνουν. Είπατε κάποια πράγματα, αν λέγατε κάτι παραπάνω θα με βοηθούσατε πάρα πολύ. Δεύτερο, στην Ελλάδα τώρα υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα, καθώς η ανεξάρτητη, το οποίο γνωρίζετε από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θεωρείται ότι φουσκώθηκαν, φούσκωσε το έλλειμμα του 2009 και προχτές η Βουλή μας αποφάσισε να συγκροτήσει Εξεταστική Επιτροπή για να ανοιχνεύσει αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για αυτά τα ελλείμματα και πού βρίσκονται. Είναι μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Το ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι αιτία αυτού του φουσκώματος ήταν το κατά πόσον οι λογαριασμοί δημοσίων επιχειρήσεων μπαίνουν στα στατιστικά στοιχεία ή όχι. Σας παρακαλώ βοηθήστε με αν έχετε εκ της και είσαστε πρόχειρος αν και σε άλλες χώρες γίνεται τέτοια μελέτη δηλαδή αν μπαίνουν τα ελλείμματα, τα προβλήματα δημοσίων επιχειρήσεων στο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης και δημιουργούνται αντίστοιχα, αντίστοιχες αλλοιώσεις, θα έλεγε κανείς, των, στατιστικών στοιχείων. Αν είστε πρόχειρος, δώστε μου σας παρακαλώ μια εμπειρία γύρω από αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Well, I'm afraid that you... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναφέρατε κάποιες ε, λεπτομέρειες ε, στις οποίες δεν μπορώ να απαντήσω. Ε, μου είπατε ότι επέκνα την Ελλάδα, αλλά είπα και θετικά πράγματα για την Ελλάδα. Μίλησα για την ανάπτυξη εργασίας ανάμεσα στην Ελστατ και τους εθνικούς στατιστικούς οργανισμούς, κάτι που βρίσκω πολύ χρήσιμο. Δύσκολο στοιχείο, και γι' αυτό στείλαμε επιστολή προς τις αρχές, βρήκαμε ότι είναι η πολύ ισχυρή πολιτική πίεση στην ανεξάρτητη στατιστική αρχή, στην Εθνική Στατιστική Αρχή και, και προς τη διεύθυνση της, ε, εθνική, της Ανεξάρτητης Εθνικής Στατιστικής Αρχής. Και αυτό το θεωρούμε αδικαιολόγητο να ασκείται πολιτική πίεση. Θεωρούμε ότι είναι προσπάθεια Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται προσπάθεια να υποβάλλονται ε, καλής ποιότητας στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα και αυτό ήταν ε, ιδιαίτερα ενοχλητικό στοιχείο για μας. Ειλικρινά, δεν μπορώ να σας ε, δώσω λεπτομέρειες για τα στοιχεία του ελλείμματος του 2009 αλλά πιστεύω ότι η συνεργασία που είδαμε και η εις συνεργασία που είδαμε ανάμεσα ιδιαίτερα στην Eurostat και τις εθνικές αρχές έχουν οδηγήσει σε μια εικόνα την οποία πρέπει να θεωρήσουμε καλή υπό τις παρούσες συνθήκες. Δεν έχω λόγους να πιστεύω ότι τα στοιχεία αυτά έχουν τροποποιηθεί με κάποιο τρόπο. και πιστεύω ότι πραγματικά υπήρξε προσπάθεια να δοθεί ακριβή εικόνα. Όσον αφορά ε, το, το φούσκωμα του χρέους, ε, φοβάμαι ότι όταν... Συχνά εξετάζουμε το χρέος υπό το φως του ΑΕΠ. Όταν έχει κανείς μια οικονομία η οποία συρρυκνώνεται γρήγορα και ταυτόχρονα να φουσκώνει ε, το χρέος του δημοσίου τομέα, με βάση ε, ε, Είδαμε μάλλον τέτοιες ε, εξελίξεις στην Ελλάδα και δεν έχω λόγους να πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ε, αποτέλεσμα λάθος στατιστικών στοιχείων. Εγώ αυτό μπορώ να το εξηγήσω κάλλιστα με όρους οικονομικής δυναμικής. Ευχαριστώ, Έτουαρτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κερχόλμ για μια πολύ ε, ξεκάθαρη παρουσίαση, για μια πολύ σαφή παρουσίαση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι στατιστικές αποτέλεσαν την πηγή της κρίσης, αλλά ε, σίγουρα άφησαν ε, να, να, κρύβεται το πρόβλημα επί πολύ καιρό και να χειροτερεύει. Είδαμε το αποτέλεσμα της περίπτωσης Lehman Brothers όταν αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία. Όταν κανείς λοιπόν μιλάει για ε, συμβουλευτικό ε, φορέα 7 ε, επίτιμων μελών σε σχέση με το κόστος της κρίσης, σίγουρα δεν υπάρχει σύγκριση. Και δεν παίρνουμε πολύ στα σοβαρά το θέμα αυτό. Αυτό αποτελεί δείγμα του τι κάνουμε σε σχέση με το τι απαιτείται. Πόσο μάλλον όταν έχουμε έναν κώδικα διοντολογία, ο οποίο θέλουμε να εφαρμοστεί απόλυτα. Όσον αφορά την ανεξαρτησία της Eurostat, ναι, ίσως να μπορούμε να περιμένουμε λίγο περισσότερο, αλλά δεν, φανταστείτε τώρα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να απαιτεί από τις, ε, να μην είναι ήδη ανεξάρτητη, ενώ ζητάει από τα, τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες να είναι ανεξάρτητες. Ε, και, ε, Μία τελευταία παρατήρηση όσον αφορά τις αποκλήσεις που δίδονται στις πολύ μικρές χώρες που δεν έχουν το απαραίτητο δυναμικό. Ε, εντάξει, διότι έτσι δεν χρειάζεται να υποβάλλονται τα απαραίτητα στοιχεία, αλλά κάθε χώρα είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει το δικαίωμα να ε, συμπεριλαμβάνεται σε διάφορες μελέτες. Δεν λύνεται λοιπόν έτσι το πρόβλημα. Οι χώρες αυτές χρειάζονται δυναμικό και εμπειρογνωμοσύνη για να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο και να δώσουν και, να μπορέσουν να δώσουν τα στοιχεία που απαιτείται από αυτές ε, άσχετα από το μέγεθος και το δυναμικό τους. Δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά. Σίγουρα μπορώ να συμφωνήσω με την παρέμβασή σας. Um, ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή στη ζήτηση. Η ερώτησή μου άπτεται των περιφερειών στις τροπολογίες μας να καταστήσουμε σαφές ότι περιμένουμε πολλά περισσότερα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις περιφέρειες. Θεωρείτε πως θα αποτελέσει πρόβλημα για το στατιστικό σύστημα. Δεν νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα για το στατιστικό σύστημα, αλλά θα είναι πρόβλημα σχετικά με την διαθεσιμότητα των πόρων. Σε μερικές περιπτώσεις, όχι μόνο στο περιφέρειες, το βλέπουμε για θέματα επενδύσεων, αλλά και άλλα ζητήματα, παρατηρούμε πως ε, υπάρχουν όλο και περισσότερα αιτήματα σχετικά με την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν κρίνουμε πως είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο αυτό να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες και ενδεχομένως να πάψουμε να κάνουμε κάποια πράγματα προκειμένου να εξοικονομήσουμε πόρους για να δώσουμε σε άλλους τομείς, σε άλλες δράσεις για να ολοκληρώσουμε μια αποτελεσματική στατική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος επιθυμεί να σε ερωτήσεις. Έχουμε μια δεύτερη ερώτηση. Έχουμε ακόμα πέντε λεπτά στη διάθεσή μας. Έχετε κάτι που σας απασχολεί. Κοιτάξτε, όταν κανεί ε, δεν έχει να πει κάτι συγκεκριμένο, καλύτερα να μην μιλήσει, διότι μπορεί να πει ανοησίε. έχουμε να συζητήσουμε το θέμα από το 2010. Εν πάση σας ευχαριστώ που βρεθήκατε σήμερα ανάμεσά μας. Πολλές θεριστικές ε, μελέτες ε, περνάνε από μπροστά μας. Εγώ χρειάζεται να τα αναγνώσω, να τις κοιτάξω, διότι κανείς δεν θα το πράξει στη θέση μου. Εν περιπτώσει, καταγράψαμε αυτά που μας είπατε σχετικά με τα προβλήματα και τους περιορισμούς που αντιμετωπίσατε με το συμβουλευτικό, στον συμβουλευτικό φορέα. Right. Well, uh, with that we... Ωραία. Έχουμε μερικά λεπτά για να στήσουμε το ESCAB 2010. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είμαι εγώ η Και θα μιλήσω από την έδρα Αρχές Δεκεμβρίου υποβλήθηκε η έκθεση και μέχρι 18 Ιανουαρίου είχατε χρόνο για την κατάθεση τροπολογιών. Ζητήσαμε επίσης και σχόλια από την Eurostat και από άλλους φορείς ε, επί της εκθέσεως. Ε, οι τροπολογίες έρχονται να κυκλοφορήσουν και ανάμεσα στους σκιώδεις συγητές. Να πω λοιπόν μερικά λόγια ευχαριστώντας όλα τα μέλη λοιπόν, που υπέβαλαν τροπολογίες. Δεν θα αφήξω τις τροπολογίες αυτές, διότι φαντάζομαι ότι τα μέλη θα το πράξουν. Παρακαλώ οι σιωπή, δεν θέλω να έχω συναγωνισμό με τους ε, ομιλούντες εντός της αθούσης. Τώρα, για τις παρεκκλήσεις, που είναι ένα ζήτημα, Φαίνεται πως μπορεί να υπάρξει συνένεση πως οι παρεκκλήσεις θα πρέπει να είναι προσωρινού χαρακτήρα προκειμένου να επιτρέψουν τα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τα ε, στατιστικά του συστήματα. Ο Έντουαρτ πρότεινε πως η Κομισιόν θα πρέπει να παρέχει πόρους και εμπειρογνωμοσύνη τα κράτη-μέλη που χρειάζονται. Ε, πρόκειται για μικρά κράτη-μέλη, διότι δεν θέλει να απουσιάζουν στοιχεία. Θα μπορείς να βρεθεί μια συμβασμός φορικά με την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. στο θέμα των περιφερειακών στατιστικών υπάρχουν πολλές τροπολογίες από τον Μοντρεμόζα. Εδώ η Eurostat ε, ανησυχεί πως αν θέσουμε κάποιους κανόνες για τις περιφέρειες, αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί και διασυνοριακά ε, κράτη-μέλη τα οποία έχουν αυτόνομες περιφερειακές κυβερνήσεις όπως ε, η Καταλωνία στην Ισπανία. Χρειάζεται λοιπόν να σκεφτούμε λίγο παραπάνω το ζήτημα και να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Η ε, γεγονός είναι ότι θέλουμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στις περιφέρειες, αλλά δεν μπορεί να βρεθεί ένα σύστημα που να ταιριάζει σε όλες. Ε, πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο να μην είναι ιδιαίτερα δυσκίνητο και χρονοβόρο και πανήρω τώρα η τροπολογία 20 και κάποιες που έχω που κατέθεσα αργότερα 36 παραδείγματος χάρη που αφορούν στο ζήτημα το κρατήριο το 50% για το κατά πόσο μια οντότητα, λογαριασμό μια οντότητα θα πρέπει να είναι δημόσια ιδιωτική. Να υπενθυμίσω εδώ ότι το 5% του κόστους καλύπτεται από πωλήσει, τότε μπορεί να θεωρηθεί ως ιδιωτική οντότητα και το σχετικό χρέος δεν μπαίνει στο πλαίσιο των κριτηρίων χρέους και ελλείμματος. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν μεγάλους οργανισμούς όπως νοσοκομεία που να ε, ε, μην περιλαμβάνονται στους ε, ισολογισμούς των κρατών μελών όπως οι ΗΠΑ Πολιτείες πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το 100% το κριτήριο 100% το πρόβλημα το οποίο μου ετέθη σχετικά είναι πως αν το πράξουμε τότε όλα τα στοιχεία χρέους και ελλείμματος θα επιδεινωθούν ε, δέχεται να υπάρξει ένα μηχανισμός ε, μέσω του οποίου να μπορούμε είτε να έχουμε τους, ε, τα στοιχεία και να τα συνδυάζουμε, τα συγκρίνουμε. Κατανοώ ότι υπάρχει ένας μηχανισμός όπου το χρέος μπορεί να αποκριθεί. αποκριθεί και αυτό δεν νομίζω ότι είναι ορθό. Γι' αυτό λοιπόν κλείνω να διατηρήσουμε το κριτήριο του 100% προκειμένου να μπορέσουμε να προοδεύσουμε. Και θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη των συναδέλφων τώρα για την υποβολή και την υποθεσμία υποβολής τροπολογία 63 να μην εξαιρεθούν ε, κράτη από τον κανόνα T85 τα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν ε, ε, πληρούν αυτών των κανόνων. Θα μπορούσαν λοιπόν να προτείνω να εξευρεθεί μια λύση με το ζήτημα αυτό. Ε, ξέρω πως η Eurostat θα ήθελε να υπάρχει ένας κανόνας για όλους, αλλά αυτό ενδεχόμενα να είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τώρα κράτη μέλη τα οποία προτίθεται να ενταχθούν στην Ευρωζώνη. Αυτό θα αφορά την προετοιμασία, θα πρέπει να επιταχύνουν κατά πέντε ημέρες, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα τα οποία χρειάζεται να πράξουν για να ενταχθούν στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι ίσονο σημασία ε, θέμα μπροστά όλα τα όσα θα χρειαστεί να κάνουν. Θα πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε λίγο παραπάνω, προτού να υποβάλουμε κάποιες συμβασικές τροπολογίες. Και τώρα με τα χαράς ε, να δώσω το λόγο στους Σκιώδης ε, εκ μέρους του ΕΛΚ ο Θέοντορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν... έχουμε πολλά προβλήματα με τις τροπολογίες. Ωστόσο, υπάρχει μία τροπολογία που έχει να κάνει με ε, τις στρατιωτικές δαπάνες, με την οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω ούτε εγώ, ούτε νομίζω οι συνάδελφοί μου. Να θεωρούνται οι στρατιωτικές δαπάνες λειτουργικές δαπάνες. θα πρέπει να μιλάμε για επενδύσεις και λειτουργικές ε, δαπάνες ε, στα πλαίσια των στρατιωτικών δαπανών, διότι αλλιώς θα είναι πολύ περίεργο να δούμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ ως λειτουργικό κόστος. Φυσικά, σε κανέναν δεν αρέσουν οι στρατιωτικές δαπάνες, οι δαπάνες άμυνας, αλλά θα πρέπει να ε, τις εξετάσουμε όπως οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της χώρας. Κατά τα άλλα, συμφωνώ απόλυτα με το υπόλοιπο της πρότασής σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Έντουαρτ. Θα είμαι κι εγώ σύντομος. Ιδιαίτερα καθότι ε, μερικά σημεία τα κάλυψα κατά την προηγούμενη συζήτηση. Να ξεκινήσω από το τελευταίο σημείο, το 100%. Δεν είναι Ε, εύκολο. Στην αρχή ήμουν αρκετά ουδέτερο, αν θα είναι 50 ή 100%. Αλλά από τεχνική άποψη ε, νομίζω ότι το 100% είναι πιο κατάλληλο ποσοστό. Όσον αφορά τις μελέτες ε, της Eurostat και του OSA στον τομέα των περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνθήκων, νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχιστούν ιδιαίτερα όταν μιλάμε για απασχόληση και πράσινες θέσεις απασχόλησης. Είναι σημαντικό οι εθνικοί λογαριασμοί να έχουν μια μορφή που να βοηθάει την διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα αυτών. Όσον αφορά το θέμα των περιφερειακών λογαριασμών, δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς εδώ. Εκτός αν κάθε χώρα επιλέξει διαφορετική μεθοδολογία υπό το φως ε, των ειδικών συνθήκων της. Όσον αφορά τις παρεκκλήσεις, παρουσίασα το επιχείρημά μου, δεν λύνουν το πρόβλημα. Ε, ε, μια χώρα μπορεί να μην έχει δυναμικό, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα της μη παροχής των στοιχείων. Και τέλος, το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων είναι κάτι το οποίο θα ελέγξω, αλλά η τροπολογία μας είχε το νόημα Εφόσον αποφασίσουμε ε, πάνω σε έναν δείκτη και κάθε χώρα γνωρίζει τι είναι αυτός ο δείκτης ή τι είναι το συγκεκριμένο σημείο αναφοράς, ε, δεν μπορεί να ε, αναθέσει μια κατοξιδότηση πράξη που να αλλάζει τη φύση αυτού του δείκτη. Το Κοινοβούλιο λαμβάνει απόφαση για το σημείο αναφοράς αυτό, το benchmark, και δεν ε, θα πρέπει να ανατεθεί σε κανέναν άλλον σχετική απόφαση. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Φίλιπ Λάμπερτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, κυρία Πρόεδρε. Έχω παρατηρήσεις για δύο τροποποίησεις που με ανησύχησαν κάπως. Ε, με ανησύχησε ο τρόπος που απαντά σε εμάς η Eurostat. Όταν εμείς υποβάλλουμε τροπολογία και η Eurostat λέει όχι, ε, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό ως απάντηση. Δεν ξέρω αν είναι κανείς παρόν από τη Eurostat, αλλά ε, θα ήθελα να επιμείνω σε δύο τροπολογίες. Η πρώτη αφορά το να λαμβάνεται το να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι από τι ε, υπηρεσίε χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Εμεί ουσιαστικά λέμε ότι η Κομισιόν μέχρι το τέλο του 2012 θα πρέπει, φέτος δηλαδή, θα πρέπει με πράξει ε, κατεξουσιοδότηση να δημιουργήσει ένα μηχανισμό για αυτού του είδου τι ε, τις και υπηρεσίε, λαμβάνοντα υπόψη μία μέθοδο που να είναι προσαρμοσμένη στον κίνδυνο. Ε, η απάντηση της Eurostat είναι ότι όχι, πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα των ε, ε, δοκιμών που γίνονται αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη μεθοδολογία. Βρίσκω πολύ σύντομη αυτή την απάντηση και εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση για να δούμε αποτελέσματα εδώ. Διότι αλλιώς μπορούμε να περιμένουμε και άλλες μελέτες, ενώ θα γνωρίζουμε ότι ο τρόπος που υπολογίζουμε τον κίνδυνο δεν αντικατοπτρίζει την δημιουργία αξίας. Ε, αυτά όσον αφορά τι γενικέ στατιστικέ. Επιμένουμε σε αυτό το θέμα δηλαδή. Ε, και η δεύτερη ε, παρατήρηση αφορά αυτή την περιβόητη έκθεση το ΑΕΠ και πέρα από αυτό. Εμείς θέλουμε εφαρμογή αυτών που ψήφισε το Κοινοβούλιο και η απάντηση της Eurostat είναι όχι. Εμείς ε, θα ε, συμπληρώνουμε το ΑΕΠ με ε, δορυφορικούς λογαριασμούς. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να υποχωρήσουμε στα δύο αυτά σημεία. Αυτές είναι οι μόνες μου παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Βίκη. Thank you. Um... Ευχαριστώ. Υποθέτω ότι κάποια από τα θέματα αυτά έχουν να κάνουν με τις αρχές που θεσπίσαμε στην οδηγία για ε, το δημοσιονομικό πλαίσιο. Στην οδηγία αυτή αναφέραμε την ανάγκη να εξεταστούν ε, τα περιφερειακά, κοινοτικά και κρατικά χρέη. Συμφωνώ όμως ότι για κάποιες περιφέρειες ε, σαν την ε, δική μου, ε, που δεν είναι αυτόνομη περιφέρεια. Δεν έχει νόημα η διαδικασία αυτή, αλλά για, για αυτόνομες περιφέρειες νομίζω θα είναι πολύ χρήσιμο κάτι τέτοιο. Θα υποβάλουμε μια πρόταση διατύπωσης. Όσον αφορά το κριτήριο του 50% και θα το θυμάται αυτό ο Φιλίπ, είχαμε μακρά συζήτηση ε, όσον αφορά την ε, κοινοποίηση ε, των ευθυνών. Δεν είμαι βέβαιη αν το 50% ή το 100% θα μας φέρουν εκεί που θέλουμε. Να καταλάβουμε δηλαδή που ε, υπάρχουν χρέη και ελλείμματα τα οποία πρέπει να, ε, ε, να κοινοποιηθούν. Αλλά δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε να τα πετύχουμε αυτά με το 50% ή 100%. Όσον αφορά τα νούμερα στην τροπολογία μου, φοβάμαι πως έχω κάνει λάθος η τροπολογία μου ε, ήθελε να αφήσουμε στις 90 μέρες ε, τα κράτη-μέλη που δεν είναι εδώ στις Ευρωζώνης και για την Ευρωζώνη να έχουμε 85 μέρες ε, και να προχωρήσουμε σε 82 μέρες. Μπορεί αυτό να ακούγεται πολύ τεχνικό, αλλά ασχολούμαστε με την σύγκριση στοιχείων από ουσιαστικά κάθε τομέα της οικονομίας μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορεί κάτι τέτοιο να στοιχήσει πολύ. Εάν τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης ε, θέλουν ε, να ε, ακολουθήσουν γρηγορότερου ρυθμού με κίνδυνο το υψηλότερο κόστος των στοιχείων, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα είναι και τόσο ακριβή τα στοιχεία αυτά. Αν θέλουν να το κάνουν αυτό, αν θέλουν να ε, ενεργήσουν πιο γρήγορα, αυτό να αποτελεί ε, επιλογή του. Αλλά ε, μου έχουν πει ότι ο κίνδυνο για άλλε χώρε μπορεί να είναι ότι αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ δαπανηρό και να είναι ει βάρο τη ακρίβεια των στοιχείων. σω λοιπόν μπορούμε να το ξανακοιτάξουμε αυτό. Και Συνεργάστηκα με τον ε, Φίλιπ σχετικά με το ε, ΑΕΠ και πέρα από το ΑΕΠ, την σχετική έκθεση. Ε, νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Αναφέρατε ότι, ότι υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει. Είναι πολύ λογική η ε, γραμμή που παρουσιάζεται. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές. Ε, θα, θα χαρώ πολύ να συζητήσουμε τα θέματα αυτά σε κάποια τεχνική συζήτηση ε, των σκιωδών εισηγητών. Ευχαριστώ. Τέλος, ο, ο Τόμας Χάντελ, παρακαλώ. δεν φαίνεται να είναι παρόν. Ωραία, ακούσαμε τους κοιόδης εισηγητές. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Και έχουμε παρόντα κάποιον από την Eurostat. Δεν ξέρω εάν θέλετε να πάρετε το λόγο. Εάν το κάνετε μπορεί να έχουμε συμπληρωματικές ερωτήσεις. Θα σας δώσω το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους σας για, την, για τις χρήσιμες παρατηρήσεις σας. Θα ήθελα να ε, απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις σας. Ε, έχουν διανεμηθεί ε, κάποιες απαντήσεις μας ε, στις ε, προτάσεις τροπολογιών. Όσον αφορά το θέμα των αποκλήσεων. Ο τρόπος με τον οποίο η Eurostat και η Κομισιόν βλέπουν τις παρεκκλήσεις είναι ότι θα πρέπει να επιτρέπουν στο εν λόγω κράτος μέλος να δημιουργήσει νέες στατιστικές πηγές, ε, μητρώα, μελέτες ώστε να μπορούν ε, έτσι να αξιολογηθούν σωστά τα στοιχεία αυτά από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δούμε τις παρεκκλήσεις σε συνδυασμό με αυτά και να μην το συνδέουμε αποκλειστικά με το θέμα των πόρων ε, και του μεγέθους. Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση. Έχουμε κάποιε μικρέ χώρε που μπορούν να υποβάλουν στοιχεία, ενώ μεγαλύτερε χώρε σε κάποιε περιπτώσει δεν μπορούν. Συμφωνούμε ότι οι παρεκκλήσει θα πρέπει να είναι προσωρινές ώστε να επιτρέψουν στη χώρα να προσαρμοστεί και πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμο εάν ο συνολικός αριθμός παρεκκλήσεων περιοριστεί ώστε η ποιότητα των στατιστικών σε ευρωπαϊκό, στοιχείο, να μην σε ευρωπαϊκό επίπεδο συγγνώμη, να μην διακυβεύεται. Ε, να διασφαλίσετε δηλαδή η συγκρισιμότητα των στοιχείων. Το δεύτερο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι το θέμα της μεταφοράς από το 50% στο 100% όσον αφορά την διάκριση ανάμεσα στους φορείς της αγοράς ε, και ε, τους ε, μη φορείς της αγοράς. Αυτό θα έχει σημαντικές συνέπειες. Έτσι θα ξεφύγουμε από την ιδέα της γενικής διακυβέρνησης στην ιδέα του δημοσίου τομέα, στον οποίο περιλαμβάνουμε στη γενική διακυβέρνηση, συμπεριλαμβάνουμε φορείς που λειτουργούν στην κανονική αγορά. Αυτό σίγουρα ε, δεν ε, εννοείται στα εθνικά συστήματα λογαριασμός. Η οικονομική ε, συμπεριφορά είναι η μέθοδος και όχι η κερδοσκοπία. Θα πρέπει να έχουμε ε, κατά νου ότι στο σχέδιο του ESA ε, ε, θέλουμε ένα συμπλήρωμα στο κριτήριο του 50%. Δηλαδή, εάν κάποια οντότητα ε, εξετάζει το κόστος της μέχρι ε, ενός ε, ύψους 50% και μπορεί να υπάρχουν κάποια ποιοτικά στοιχεία τα οποία να δείχνουν ότι η οντότητα αυτή δεν ανήκει στην αγορά, μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε non-market. Επίσης, ε, στην ε, συνθήκη του Μάστριχ μιλάμε για ε, γενική διακυβέρνηση και όχι για δημόσιο τομέα. Αναγνωρίζουμε την χρησιμότητα ενός μηχανισμού με τον οποίο... Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, δεν ακούω και θα ήθελα πολύ να ακούσω την παρέμβαση του κυρίου. Ε, πολλοί μιλούν εδώ πίσω. Ναι, εγώ έβαλα τα ακουστικά μου για να μην ακούω. Ε, ομιλητής. Ε, θα αναφερθώ πάλι στο θέμα της μετακίνηση από το 50% στο 100%. Να σας πω απλά ότι στην συνθήκη του Μάστριχτ αναφερόμαστε στη γενική διακυβέρνηση και όχι στον δημόσιο τομέα. Θα θεωρούμε χρήσιμο όμως να υπάρχει ένας μηχανισμός όπου θα έχουμε μια πλήρη σειρά στατιστικών στοιχείων και ε, αν είναι απαραίτητο μπορούμε να δώσουμε στοιχεία για το δημόσιο τομέα ως πρόσθετες πληροφορίες. Επίσης, αναφέρθηκε το θέμα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και το θέμα του κινδύνου. Στην παρούσα ESA του 2010, η συμφωνία που ε, επιτέθηκε από τους Ευρωπαίους ε, Εμπειρογνώμονες ε, ήταν να λέμε ότι η χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση συνεπάγεται ότι θέτει κανείς τον εαυτό του σε κίνδυνο. Γι' αυτό η αμοιβή αυτού του κινδύνου θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις εκροές όσον αφορά την διαμεσολάβηση και γι' αυτό ο κίνδυνος συμπεριλαμβάνεται εδώ. σε μια κρίσιμη κατάσταση, σε μια κατάσταση κρίσης όπου ε, υπάρχει μεγάλη αστάθεια στις αγορές, συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί μια task force, μια ειδική ομάδα η οποία θα εξετάσει ποια θα είναι τα αποτελέσματα εάν αποκλείσουμε τον κίνδυνο. Και περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτή τη task force, αυτή τη ε, ειδική ομάδα, ε, που θα μα εξηγήσει τι σημαίνει αυτό όσον αφορά τη μεθοδολογία. Η ομάδα αυτή έχει ολοκληρώσει τι εργασίε τη. Τον Ιούνιο θα ε, συζητηθεί, ε, θα συζητηθούν αποτελέσματα από την ε, CMFP, την Αρμόδια Επιτροπή και εάν προκύψει από εκεί μια πιο ισχυρή μεθοδολογία θα μπορέσουμε να την συμπεριλάβουμε στην ESA 2010. Αλλά και πάλι η συμφωνία μεταξύ του μεγαλύτερου μέρους των εμπειρογνωμόνων ήταν ότι εάν ε, δεν ε, διακινδυνεύσει κανεί, ε, ουσιαστικά δεν κάνει χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Και μετά υπάρχει το θέμα τη έκθεση GTB and Beyond, ΑΕΠ και πέρα από το ΑΕΠ. Σε αυτήν την φάση των άτυπων ανταλλαγών δεν είμαστε υπέρ αυτού. Η θέση μας είναι να λέμε ότι θα θέλαμε να συμπληρώσουμε το ΑΕΠ με κάποιους δορυφορικούς λογαριασμούς. Αυτή η δορυφορική ε, λογαριασμοί επιτρέπουν να έχουμε κάποιους νομισματικούς και μη νομισματικούς δείκτες. Θέλουμε να έχουμε μια ευρεία, πλήρη βάση για τη λήψη αποφάσεων. Και αυτοί οι δορυφορικοί λογαριασμοί είναι πολύ ακριβείς, ιδιαίτερα όσον αφορά το περιβάλλον. Υπάρχει ένα ε, διεθνές πλαίσιο λογαριασμών και υπάρχει και κανονισμός ευρωπαϊκός που ρυθμίζει αυτούς ε, τους δορυφορικούς λογαριασμούς. Ε, και είναι πολύ καλός τρόπος εργασίας αυτός. Όλοι ξέρουμε ότι ε, το θέμα της αξιολόγησης είναι πολύ δύσκολο θέμα. Άλλωστε υπάρχει και το θέμα της σχέσης της γενιάς μας με τις επόμενες γενιές που θα ε, αντίκυνται στο θέμα της ε, αξίας ε, στην αγορά. Αυτή ακριβώς είναι η καρδιά του προβλήματος ε, και γι' αυτό πιστεύω ότι μία ε, προσέγγιση που χρησιμοποιεί αυτούς τους δευτερεύοντες λογαριασμούς είναι κατάλληλη. Υπάρχει και το θέμα της περιφερειοποίησης. Όπως είπε η Πρόεδρος, ε, θα πρέπει να ε, γίνει περισσότερη δουλειά εδώ πέρα. Η Κομισιόν θέλει να ε, διασφαλίσει την δίκαιη αντιμετώπιση όλων των περιφερειών άσχετα από την θέση τους. Δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά επαχθές το όλο εγχείρημα Λόγω της ε, παρούσας ε, κατάστασης ε, των στατιστικών πόρων είναι δυνατόν να εξεταστούν οι περιφερειακοί λογαριασμοί χωρίς παραπομπή στους εθνικούς λογαριασμούς. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειαζόμαστε τεχνολογίες εχμής για να περιφερειοποιήσουμε τα στοιχεία σε εθνικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας σε διάφορες υποθέσεις. Όσον αφορά το θέμα του τι συν 85, θα πρέπει να σας πω ότι η Κομισιόν αυτή τη στιγμή πρότιμα να μείνει στη θέση της ε, τα στοιχεία αυτά, τα T 85, ε, να ε, ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη, διότι πιστεύουμε ότι Στόχο είναι στο πρόγραμμα να έχουμε ε, και το βλέμμα προς το μέλλον. Όσον αφορά τις ε, δαπάνες για την άμυνα, συμφωνούμε με αυτό που υπόθηκε νωρίτερα, ότι θα πρέπει μέρος τους ε, να θεωρηθούν τεχνικές, ενώ το άλλο μέρος να χωριστούν σε τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες. διότι μιλάμε για υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται σε μακρύ χρονικό διάστημα και αυτός άλλωστε είναι ο ορισμός του περιουσικού στοιχείου στο όλο σύστημα αυτό. Κυρία Πρόεδρε, ελπίζω να απάντησα στα θέματα που τέθηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ήταν νομίζω πολύ χρήσιμα αυτά. Οι συζητήσει αυτέ μα προωθούν περισσότερο προ την οδό που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Άκουσα τι είπε ε, ο Εντουάρτ για τι καταξιοδότηση πράξης ε, και είπε ότι ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον θα υπάρχει αυτή η εξισοδότηση για κάποιες πράξεις που δεν επιτρέπεται να, να ε, τύχουν αυτή τη μεταχείρισει. Θα το γράψουμε σαν απαγόρευση ή τι θα κάνουμε. Θα πρέπει να το δούμε για το μέλλον αυτό. Μπορώ να δεχτώ τις αρχές των όσων είπατε. Ίσως με την ε, μεθοδολογία και τις της πράξεις να μπορούσαμε να καταλήξουμε κάπου. Για τις 90 ημέρες, 82 ημέρες, μπορώ να δεχθώ το επιχείρημα της Βίκης. Γιατί να διακυβεύσουμε την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων όταν δεν υπάρχει κάποιο χρήσιμο αντιστάθεσμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει μια διευθυντική προθεσμία. Και πρέπει να υπολογίσουμε το χρόνο που περνάει μέσα στο δικό του σύστημα, ένα μήνα δηλαδή νωρίτερα. Πράγμα που είναι προς όφελος της Ευρωζώνης. Άκουσα τι είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωστάτ ότι κάποιος μηχανισμός για πλήρη εικόνα ημερομηνιών που θα οδηγεί σε δημοσίευση 100% κάτι θα πρέπει να μπορεί να γίνει, όπως είπε και η Βίκη, ίσως και κάποια άλλα πράγματα θα πρέπει να εξετάσουμε. Ή, μάλλον θα πρέπει να εργαστούμε λιγάκι περισσότερο πάνω σε αυτό το τομέα, για να ξέρουμε τι θέλουμε να επιτύχουμε. Δηλαδή να ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι ευθύνες που σχετίζονται εδώ Κάποια παρουσίαση λοιπόν. Είναι καλή. Και θα ήταν πολύ αντιφατικό να προσπαθήσουμε να ε, αλλάξουμε κριτήρια που γνωρίζουμε καλά και που έχουμε συνηθίσει. Ίσως στο μέλλον αποφασίσουμε να αλλάξουμε τα κριτήρια αυτά, αλλά προς το παρόν ας ε, αρκεστούμε στο να προχωρούμε βήμα προς βήμα. υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που θα πρέπει ακόμα να μελετηθούν όσον αφορά αυτό το θέμα των δορυφορικών λογαριασμών. Ευχαριστώ πάντως όλους εκείνους που συνέβαλαν. Τι κάνουμε τώρα? Α, θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 20 Μαρτίου και να περάσουμε στην Ολομέλεια στην πρώτη Ολομέλεια του Μαΐου. Και θα αρχίσουμε να εργάζομαι στις συμβαστικές τροπολογίες με τη βοήθεια της ε, γραμματείας των σκιωδών λίγο πολύ αμέσως. Λοιπόν, τώρα θα δώσω την προεδρία στην άλλη για τα επόμενα 45 λεπτά περίπου. Συνεχίζουμε με τη σε διάταξη. Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση του κυρίου Κάζα για διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωση. Ο εισηγητή έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον έχουμε διαρμηνία από τα Μαλτέζικα. Φαίνεται όμω όχι. Θα αναγκαστώ λοιπόν να μιλήσω αγγλικά. Ούτε πολωνικά, πολωνική διερμηνία έχουμε. Α, όχι, έχουμε διερμηνία, αλλά δεν έχουμε μέλη. Αλλά για τρίτη φορά, τονίζω, φέτος δεν έχουμε διερμηνία από και προς τα Μαλτέζικα. Την επόμενη φορά ελπίζω να έχουμε Μαλτέζικη διερμηνία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνέβαλαν στην έκθεσή μου. για εκείνους που επέβαλαν όλες τις τροπολογίες που πήρα. Δεν υπάρχουν πολλά αντιφατικά στοιχεία νομίζω σε αυτή την έκθεση. Δεν θα σπαταλήσω λοιπόν πολύ χρόνο. Καταρχήν θα ήθελα να συζητήσω τη σκέψη για την υποβολή των δικών μου συμπληρωματικών τροπολογιών Ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό είναι ότι λίγο χρόνο μετά που υπευλήθη η έκθεσή μου, πήραμε τη γνωμοδότηση της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, Προστασίας ε, Στοιχείων που ζήτησαν κάποιες τροπολογίες για να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων τη χάνει βασμό. Αυτές λοιπόν οι πραγματικές ε, τροπολογίες ευθυγραμμίζουν η έκθεση πλήρω με τις συστάσει του Υπηρεσία Εποπτεία των Ευρωπαϊκών Στοιχείων. οι φίλοι ζήτησαν να υπάρχει ένα βήμα για τους ειδικούς όρους κατανάλωσης και τον ΦΠΑ. Αντί για το λεγόμενο JPDF. Ίσως όμως αυτό να μην αρμόζει σε αυτή την έκθεση. Παρ' όλα αυτά, ίσως είναι καλό να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα ότι το Κοινοβούλιο δηλαδή είναι υπέρ της εγκαθίδρυσης ενός τέτοιου βήματο και θα ήθελα να το εφαρμόσει το γλυκορότερο δυνατόν. Θα σημειώσατε ότι συστήνω υπερψήφιση της μεγάλης πλειοψηφίας των τροπολογιών, εκ των οποίων οι περισσότερες νομίζω διευκρινίζουν το κείμενο και το εμπλουτίζουν. 8, 14, 9, 19, 30, 31, 33 36 και 41, 42. Εγώ δεν συμφωνώ με την εισαγωγή κυρώσεων, κυρίως γιατί οι περισσότερες διατάξεις αυτή τη ε, νομοθεσία είναι εθελοντικέ. και είναι αρκετό να μην υπάρχει σωστή συνεργασία σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση. Λοιπόν, προσβλέπω στι συμβολέ των συναδέλφων εδώ και ελπίζω να υιοθετηθεί με μεγάλη πλειοψηφία τελικά η εκθεσία. Με ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, και εγώ, η Σκιώδη, ο κύριο Σπούλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Κάζα για την συνεργασία πάνω σε αυτή την έκθεση. Νομίζω πετύχαμε και πολλές σημαντικές ε, αλλαγές. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε περί τίνος πρόκειται. Ενημέρωση των κανόνων, δηλαδή πιο διαφανείς κανόνες και να μπορούμε με ηλεκτρονικά μέσα να ανταλλάσσουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες. Αυτό σε γενικές γραμμές σημαίνει ότι θα αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα χωρίς να αυξήσουμε το κόστος. Και ε, τελευταία αναλύση, ε, αυτό είναι προς συμφέρον και ημών και των ε, άμεσα ενδιαφερομένων. Η ανάγκη για περισσότερο εμπιστοσύνη και συνεργασία είναι ο στόχος της νομοθεσίας. Όλες οι σημαντικές ε, πληροφορίες από τρίτες χώρες θα πρέπει επίσης να ε, μοιράζονται και με όλες τις ε, ενδιαφερόμενες χώρες. Γενικά μπορούμε να δεχτούμε την έκθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριο Σμιτ. Ευχαριστώ Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομο. Πολύ καλή έκθεση αυτή κατά τη γνώμη μου. Εργαστήκαμε πολύ στενά πετύχανε ευρεία συνένεση και ελπίζουμε θα πετύχουμε και ευρεία πλειοψηφία. Όπως είπε και ο κύριος Κάσα, για την τροπολογία 40, για ένα κοινό βήμα, νομίζω ότι το συζητήσαμε αυτό ήδη, πρέπει να είμαστε πολύ περιοριστικοί βέβαια, να είμαστε πιο γενικοί, Αλλά ελπίζω ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε συνέντευξη γιατί νομίζω θα μπορούσε να ήταν χρήσιμο. Συμπεριλαμβανομένου και του ΒΠΑ ενδεχομένω. Κάποια σχόλια για τις άλλες τροπολογίε. Θα μπορούσα να φανταστώ ότι η δική μου τροπολογία υπαριθμών 29 είναι εκείνη στην οποία αναφερθήκατε όσον αφορά την ε, προστασία των δεδομένων. Είναι κάπως σύντομα τα χρονικά διαστήματα. τι μπορούμε εδώ να αλλάξουμε δηλαδή την νομοθεσία. Η δική σας τροπολογία είναι κάπως ασαφής. Πρέπει να το παραδεχθείτε νομίζω. Ασαφής όσον αφορά τα χρονικά όρια. λέει κάτι επαρκής χρόνος, κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να είμαστε καλοί στους καλούς και κακοί στους κακούς νομίζω. Και κάτι πολύ λεπτό, μια που και με την ε, διαρμηνία. Έχουμε και την μετάφραση των κειμένων. Και αυτό αφορά η δική μου τροπολογία 30. θα υπάρχει νομίζω συμπληρωματικό διοικητικό κόστος εάν οι αρχές πρέπει να μεταφράζουν τα πάντα. Τι να σας πω τώρα. Τολμή, τολμώ να το πω μετά από τις δικές σας παρατηρήσεις και τη διαρμηνία προηγουμένως. Και θα ήθελα επίσης να υποστηρίξω την τροπολογία αυτό 1. την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών για να μην υπάρχει φοροδιαφυγή. 41 του κυρίου Λάμπερτς. Μπορούμε νομίζω να την υποστηρίξουμε και αυτή. Γενικά είναι καλή η έκθεση αυτή και ελπίζω να έχουμε ευρεία συνένεση. Ευχαριστώ κύριο Λάμπερτς. Well. Ah, you've got different guises. Είστε Είστε μεταφυ... Είσαστε μεταφυσμένοι Σάρον Sharon Δεν ξέρω πώς να το πω στα Μαλτέζικα, αλλά σας ε, ευχαριστώ που υιοθετήσατε τις ε, τροπολογίες μας. Τι να πω, νομίζω ότι είναι καλή η έκθεση αυτή και ότι θα έχει ευρεία υποστήριξη. Να πω στον Όλε ότι συμφωνούμε και την ε, συμφωνούμε και με, την τροπολογία σας ε, για το κοινοφόρουμ. Δεν έχουμε υποβάλει πολλές τροπολογίες, ε, διότι έχουμε περιορισμένο δυναμικό και ξέρετε ότι έχουμε κάποια σοβαρά θέματα αυτή τη στιγμή. Ε, αλλά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ισχύει ότι αν ε, το Κοινοβούλιο μπορεί να ε, στείλει ένα ισχυρό μήνυμα, δεν αποφασίζουμε σε αυτά τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι αυξάνεται έτσι η ε, δυνατότητά μας να ακουστούμε, ιδιαίτερα σε έναν τομέα πολιτικά πολύ ευαίσθητα. Μπορεί, μπορούμε να δείξουμε ότι σπρώχνουμε την Ευρώπη να προχωρήσει στα θέματα αυτά. Νομίζω ότι βοηθάει. Βλέπω λοιπόν την έκθεση αυτή ως μέρος του μηνύματός μας αυτού και συνδέεται και με την ε, έκθεση, την πρώτη ε, ετήσια φορολογική έκθεση. Ευχαριστώ. Ο, ο κύριος Φόξ. Controversial draft. And we also support the majority of the amendments tabled by the rapporteur. Είδαμε τις τροπολογίες του εισηγητή και των υπολείπων μελών. Θα ήθελα να αναφερθώ στα Τροπολογία 19 του κ. Λάμπερτ. Να πω ότι προτιμώ το αρχικό κείμενο τη Κομισιόν. Θεωρώ ότι οι αρμόδιες αρχές είναι αυτές που θα αποφασίζουν κατά πόσον απαιτείται διοικητική έρευνα και θα πρέπει να ενημερώνει αμέσω την ετούσα αρχή σε περίπτωση που δεν είναι απαραίτητη αυτή η διοικητική έρευνα. Επίσης θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα υποβολής έκθεσης, ε, να μην υποβάλουν μόνο και την έκθεση, εάν κρίνουν ότι είναι της νόμου το όφελος. Ε, τα άρθρα 23, το τροπολογή 23 του κ. Μάρτιν δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ένας πίνακας κυρώσεων για μη συμμόρφωση. Η μη συμμόρφωση θα πρέπει να ε, καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Ευχαριστούμε τον κύριο Κάσα. Πιστεύουμε ότι η έκθεσή του δεν είναι επίμαχη. Θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημά σας ε, γιατί δεν μπορείτε να μιλήσετε τη γλώσσα σας φυσικά είναι δικαίωμά σας αλλά σύμφωνα με την εκπεριτροφή της εκπεριτροπής έχουμε σήμερα με μικρότερη αίθουσα που διαθέτει 12 διερμηνευτικούς θαλαμίσκους ε, και έτσι αναγκαστικά λόγω αυτής της ε, περιτροπής και επειδή τα, ε, τα πρόσωπα τα οποία έχουν ταλέντο στις ε, γλώσσες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα, μπορείτε να εκφραστείτε άψογα σε μια άλλη γλώσσα πριν την μητρική σας, αλλά αυτός δεν είναι φυσικά λόγος να μην έχουμε και διερμηνία προς τη γλώσσα σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν έχω άλλα σχόλια να προσθέσω. Ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους μου για την υποστήριξη και σχετικά με την μαλτέζικη γλώσσα. Την επόμενη φορά θα φροντίσω να μιλήσω κινέζικα και θα δω πώς ε, θα τα βγάλετε πέρα. Εντάξει, κατανοώ το πρόβλημα, αστιεύουμε φυσικά. Δεν ε, ήθελα να επικρίνω εσάς, Πρόεδρε, απλά τα σχόλιά μου τα απευθύνονταν μάλλον στην πρόεδρο της Επιτροπής, η οποία όμως ε, δεν απάντησε στο ε, αίτημά μου. Ελπίζω λοιπόν την προσεχή φορά να έχω στη διάθεσή μου την γλώσσα και θα είμαι σε καλύτερη θέση να εξηγήσω τις θέσεις μου και τις απόψεις μου. Πάντως κάνατε εξαιρετική δουλειά, παρατηρεί η Πρόεδρος. Ε, θα ψηφίσουμε αύριο επί των 35 τροπολογιών, αύριο το πρωί.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 Να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Πρόκειται την έκθεση του κυρίου Σλάβη Μπίνευ για την επέκταση τη γεωγραφική έκταση των εργασιών της Ευρωπαϊκή Τράπεζα ε, Ανασυγκρότησης στην Νότια και Ανατολική Μεσόγειο. Και εδώ έχουμε το αυτό πρόβλημα. Α, όχι, όχι, έχουμε, έχουμε. Αποκτήσαμε, δεν είχαμε, αλλά αποκτήσαμε. Μπορείτε να αρχίσετε λοιπόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία που φρόντισε για την διαρμηνία. Η έκθεση είναι τεχνικού χαρακτήρα και καλύτερα να μπορέσω να μιλήσω την μητρική μου γλώσσα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ΕΤΕΑ συστάθηκε προκειμένου να βοηθήσει τις χώρες και αρχικά προβλέπεται να λειτουργήσει σε χώρες της πρώην ε, του Ανατολικού Μπλοκ μεταξύ αυτών και της δικής μου. Αυτά τα κράτη ε, στηρίχθηκαν προκειμένου να μεταβούν από την ε, αρχική κατάσταση της οικονομίας τους σε οικονομία της αγοράς. και οι χώρες αυτές ε, πέθησαν ε, τα τρία αλφα, τα τρία αποθητά α. Η ΕΤΑ στηρίζει προγράμματα, ενισχύει την απασχόληση και ενισχύει την ανάπτυξη σε ποικίλου ε, κλάδους. Είναι μια πολύ διαφορετική τράπεζα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Γιατί ε, μολονότι πολύ τις ε, μπλέκουν θα έλεγα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει περισσότερο γεωπολιτικό ρόλο και έναν ευρύτερο στόχο. Ενώ η ΕΤΕΑ στηρίζει τον ιδιωτικό τομέα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, τα χρήματά της φτάνουν σε πολύ περισσότερους ε, ανθρώπους και τα δύο θεσμικά όργανα ασχολούνται με τον αυτό στόχο αλλά συνεργάζονται και δεν ε, δημιουργούν επικαλύψεις. Ιδιαίτερα σε περιπτώσει όπου υπάρχει κάποια διαφορά. Τώρα, οι τροπολογίες ε, αφορούν ε, τις χώρες ε, της κεντρικής και νοτίου Ευρώπης Γιατί λοιπόν συζητάμε την έκθεση αυτή τώρα, διότι το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να καταδείξει πως στηρίζει τις ε, διαδικασίες ε, που έχουν ξεκινήσει στην ε, Βόρειο Αφρική μετά από την Αραβική Ένωση, Άνοιξη και θα πρέπει να δείξουμε πως είμαστε έτοιμοι να δράσουμε, να ενεργήσουμε για τις, στις χώρες αυτές. Αυτό είναι σημαντικό να συμβεί τώρα, διότι αυτή είναι η σωστή στιγμή που οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να προωθηθούν. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αντανακλάται στα προγράμματα που προωθεί η τράπεζα και ε, φυσικά θα χρησιμοποιηθούν πόροι της ε, τράπεζας ε, ανεξάρτητα από τα ποσά τα οποία έχουν δεσμευθεί από άλλους ε, θεσμούς και Ούτε εδώ λοιπόν θα υπάρξει επικάλυψη διότι και επιπλέον η τράπεζα θα χρησιμοποιήσει μια νέα προσέγγιση για τα νέα κράτη. Τώρα αναφορικά με την ασφάλεια, την εφαρμογή των προγραμμάτων, ε, τα και για να να εφαρμοστούν το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκή Τράπεζα ανάπτυξη και Ανασυγκρότησης ε, θα υπάρξει παρακολούθηση, αποκτία με όργανα τα οποία ήδη λειτουργούν επιτοπίω ε, και αν δεν πληρούνται τα πολιτικά κριτήρια τότε η τράπεζα δεν θα χορηγεί τους ε, πόρους. Λοιπόν, ε, θα γίνεται η κατάλληλη παρακολούθηση, το πού πηγαίνουν τα χρήματα, προκειμένου να μην υπάρχει εκτροπή αυτών. Οι εμπειρογνώμονες ε, θα μεταβούν επιτόπου, προκειμένου να αξιολογήσουν ε, την, στην κατάσταση, την, πώς έχει η διαφθορά η τράπεζα θα συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη των ε, περιοχών. Οι επενδύσεις ε, δεν ε, θα εστιάσουν στα ορυκτά καύσιμα. Του αντίον στόχος είναι η ενέργεια με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. και ο τομέας ενέργειας ε, καλύπτει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό από, τον, ε, από τα κονδύλια τα οποία χορηγούνται. Το, τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ε, ιδιαίτερη σημασία για την ΕΤΑ. Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική της τράπεζας για την στήριξη των πληθυσμών, την ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση της ένδυας κλπ. Εάν υπάρξουν προβλήματα τότε θα διακοπούν οι χρηματοδοτήσεις. 20 κράτη πληρούν ε, τα κριτήρια του ΠΟΕ και ε, προωθούν την οικονομία της αγοράς. Ε, υπάρχει διαφάνεια από πλευράς ΕΤΑ διότι υπάρχουν αιτήσεις εκθέσεις ε, σχετικά με την ε, λειτουργία της τράπεζας ε, στις περιοχές αυτές. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να επιταχύνουμε τις διαδικασίες διότι έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πανέτοιμο να υποστηρίξει τέτοιες προσπάθειες όχι μόνο με λόγια αλλά και στην πράξη για τον περαιτέρω και δημοκρατισμό των χωρών αυτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα τις παρατηρήσεις ε, των ε, σκιωδών εισηγητών. Ε, πρώτα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να κάνω την παρατήρηση ότι δεν υπάρχει διερμηνία προς τα φιλανδικά. Φαίνεται όμως ότι και εμείς είμαστε ιδιαίτερα γλωσσομαθείς. Καταρχήν θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι επικροτώ την ε, πρόταση για ε, την επέκταση του ΕΤΑ στην ε, Νότια και Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα τα οποία πιστεύω ότι θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στα, στις τροπολογίες. Πιστεύω ότι θα πρέπει οι χώρες στις οποίες ενεργοποιείται η ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την ε, Ανάπτυξη να πρέπει να πληρούν ε, διάφορε διάφορες προϋποθέσεις. Θα πρέπει να είναι διατεθειμένες να ακολουθήσουν τις αρχές της δημοκρατίας του κράτους δικαίου, να σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως είναι το, η ελευθερία της έκφρασης και, η ανεξιθρησκεία. Ο ρόλος ακραίων Ισλαμιστικών κομμάτων ε, μπορεί να απειλούν ε, ε, κάποια βασικά θεμελιώδη δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη θα πρέπει να ακολουθεί την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Καλής Γειτονίας η σχετική αναθεώρηση θα καλύψει ε, πέντε βασικά ε, στοιχεία. Τις ελεύθερες δίκαιες εκλογές, ε, την ελευθερία έκφρασης του συνέρχεστε και την ελευθερία της, του τύπου, κράτος δικαίου, δημοκρατικό έλεγχο στην άμυνα στις δυνάμεις. Η θέση ε, των χωρών της ε, Νότιας Μεσογείου όσον αφορά την ε, διακυβέρνηση, την διαφθορά και τα λοιπά. Μετά την Αραβική Άνοιξη θα πρέπει να επικεντρωθεί ιδιαίτερα σε αυτές τις χώρες η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη. Αποτελεί ευθύνη της OCCO να ασχολείται με θέματα κεραιότητας, ε, λογοδοσίας, ε, ε, την καταπολέμηση της, της τρομοκρατίας και άλλα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης έχει επικριθεί. Ελπίζω όμως ότι ο συντονισμός των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη με άλλους φορείς θα ενισχυθεί ώστε να αποφύγουμε επικάλυψη εργασιών και να μπορέσουν τα διάφορα μέτρα να είναι ε, συνεπή και να στηρίζουν το ένα το άλλο. Ε, ακούστηκαν και επικρίσεις όσον αφορά τα προγράμματα ενέργειας που έχει στηρίξει η ΕΤΑ. Πιστεύω ότι οι χώρες της Ανατολικής και Νοτιού Μεσογείου ε, έχουν μια μοναδική ευκαιρία να προωθήσουν προγράμματα βιώσιμης ενέργειας. Ε, μπορούσαν να συμπεριληφθούν και άλλα ε, πράγματα στα εκτιμώντα. Ε, Προσλέπω όμω στην καλή συνεργασία με τον εισηγητή, καθώ και με του άλλου εισηγητέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κούτα, παρακαλώ. Salut și Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ επικροτώ την πρόταση για την διεύρυνση ε, των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ε, στη Μεσόγειο. Και χαίρομαι που ο εισηγητής ε, συμφωνεί και αυτός με την πρόταση αυτή. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη έκθεση, μια έκθεση με συνεκτικότητα, ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά που η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει δηλώσει επανειλημμένα σε διακηρύξεις ε, και που αφορούν ε, τις αραβικές χώρες στη Μεσόγειο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης έχει μακρόχρονη πείρα στον τομέα αυτών και Ελπίζω να συμμετάσχει στη ε, μετάβαση στη δημοκρατία των ε, χωρών των χωρών ε, που πριν ήταν κομμουνιστικές. Και αυτό πιστεύω θα πρέπει να το περιλάβουμε και θα ήθελα να αναφερθώ και στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών αυτών. Η οικονομική ανάπτυξή τους θα πρέπει να στηριχθεί επίση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και ανάπτυξη. Θα ήθελα να εκφράσω και την πεποίθησή μου ότι μαζί με τους και ε, εισηγητές θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ε, πολύ καλή έκθεση και είμαι διατεθειμένος ε, να συμβάλλω σε αυτήν. Ευχαριστώ κύριος Λάμπερτς, παρακαλώ. Ε, έχω διερμηνεί από τη γλώσσα μου, αλλά ε, σεβόμενος τους συναδέλφους ε, θα μιλήσω στα αγγλικά, ώστε να μην χρειάζεται ε, να φορέσετε ακουστικά. μπορώ να συμφωνήσω με πολλά από όσα είπες. δεν θα τα αναπτύξω περαιτέρω. Η, η απόδοση... Η, η, οι δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη στον τομέα τη ενέργεια ε, δεν είναι κάτι το οποίο ε, μα βρίσκει συμφώνου. Ε, Παρεπιπτόντω και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεω ναι, υπόκειται στι ίδιε επικρίσει. Επίση, συμφωνώ με διάφορα άλλα που είπε εάν ε, διευρύνουμε την ε, εντολή της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, δεν συνδέεται αυτό άμεσα με την με τις ερήτρες περί δημοκρατίας αλλά υπάρχουν χώρες που δεν πληρούν τα κριτήρια περί δημοκρατίας, η Ρωσία, το Καζακστάν κτλ. Και δεν συμφωνώ να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε ενιαία μέτρα και σταθμά, αυτά που αναφέρεις και εσύ, ε, όχι όμως αυτά των νοτιών χωρών. Ε, τρίτον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης λέει ότι ε, όλοι θα πλουτίσουμε ε, και θα ε, μπορέσουμε να βγάλουμε τον κόσμο από την φτώχεια. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Η ΕΤΑ δείχνει ότι οι παρεμβάσεις πράγματι μειώνουν την φτώχεια και την ένδυα στις χώρες όπου λειτουργεί. Ένα τελευταίο θέμα. Είναι θεσμικό. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα για την Αραβική Άνοιξη. Είναι πολύ δύσκολο να πει κανεί, όχι, να μην το κάνουμε αυτό. Έτσι, ε, ε, φτάνουμε σε κάπω αυτά είναι τα συμπεράσματα. Όταν ε, δημιουργούνται θεσμοί, είναι πολύ δύσκολο να καταργηθούν όταν πια δεν είναι χρήσιμοι. Το, το ΕΤΑ δημιουργήθηκε, η, ΕΤΑ δημιουργήθηκε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Εμεί πιστεύουμε ότι δεν είναι πια χρήσιμη και σε προηγούμενη έκθεση προτείναμε να συγχωνευτούν οι δραστηριότητε τη να αποτελέσει μέρο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχουμε την Αραβική Άνοιξη και ακούμε ε, ε, και από διαφόρους ε, ενδιαφερόμενους που λένε γιατί να χρησιμοποιήσουμε το μέσο αυτό για να στηρίξουμε την Αραβική Άνοιξη. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε ας αλλάξουμε την εντολή όχι να διαβρύνουμε, να αλλάξουμε την ε, εντολή της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξης και να την κάνουμε την Τράπεζα της Αραβικής ε, Άνοιξης, αλλά να φροντίσουμε να μην μπλέκεται πια σε ευρωπαϊκές υποθέσεις, όπου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να είναι ο μοναδικός φορέας. Και επίσης, μήπως η Παγκόσμια Τράπεζα μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις Αραβικής Άνοιξης. Χρειαζόμαστε πράγματι άλλο φορέα που να το κάνει αυτό. Εγώ θα προτιμούσα εξορθολογισμό να πούμε ε, η Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων να ασχοληθεί με τα ευρωπαϊκά θέματα και για θέματα όπως είναι η ε, Αραβική Άνοιξη και επειδή τα λέει ο Ομπάμα τώρα όλα αυτά δεν μπορεί όλα αυτά να τα κάνει η Παγκόσμια Τράπεζα. Εγώ θα ήθελα να εξετάσουμε εναλλακτικέ λύσει προτού να καταλήξουμε στο συμπέρασμα βιαστικά ότι έχουμε εδώ ένα θεσμικό όργανο, το οποίο δεν έχει και πάρα πολύ δουλειά. Α του δώσουμε λοιπόν λίγη δουλειά, ώστε να δικαιολογεί την ύπαρξή του. Ε, και πάλι ζούμε σε εποχέ κρίση, σε εποχέ λιτότητα και ε, η τροποποίηση αυτού του θεσμικού οργάνου για μένα, αυτή τη υπηρεσία, δεν στέλνει κατά τη γνώμη μου το σωστό μήνυμα προ τον κόσμο. Μπορεί να είναι εξορθολογισμός ο οποίος δεν βλάπτει κανέναν ε, πολίτη, αλλά ε, αφορά κάποια θεσμικά όργανα τα οποία θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Προτού λοιπόν καταλήξουμε βιαστικά στο συμπέρασμα ότι ναι, ναι, ας, ε, δώσουμε αυτή την εντολή στο όργανο αυτό ώστε να επιβιώσει, θα ήθελα πάρα πολύ να εξετάσουμε τις εναλλακτικέ λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος Καμά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αρχικά μου άρεσε πολύ η έκθεση. Επικροτώ την ε, ε, πρόταση να ε, διευρύνουμε την γεωγραφική εντολή. Θέλουμε να φαίνεται πώς κάνουμε δουλειά και όπως είπατε πολύ σωστά όσον αφορά την Αραβική Άνοιξη θέλουμε να φαίνεται ότι υποστηρίζουμε τις νέες δημοκρατίες και όταν ήμουν εισηγητή για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συμπεριλάβαμε κάποιε τροπολογίε, ώστε να είναι σαφέ ότι απλά ε, στηρίζουμε τη μετάβαση των χωρών αυτών προ την ε, ε, δημοκρατία και να μην θεωρήσουμε ότι μόνο και μόνο λόγω εραυκή άνοιξη ξαφνικά θα έχουμε δημοκρατικέ και ανοιχτέ κοινωνίε. Και θέλαμε επίση να βρούμε την σωστή ισορροπία όσον αφορά την παρέμβαση στα ιστορικά μια χώρα. Υπάρχουν ε, ε, ε, νέες δημοκρατίες στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. αυτά αφορούν ανθρώπους, και ανθρώπους που ζουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ε, είχαμε ήδη πει τότε μαζί με του αισιόδη εισηγητέ ε, για την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ε, συντονίζει τι δραστηριότητε τη με αυτήν τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη. Άκουσα αυτά που είπε ο κύριο Λάμπερτ όσον αφορά αυτό το θεσμικό όργανο και νομίζω ότι είναι σωστό το επιχείρημά του. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε μήπω έχουμε εδώ δύο θεσμικά όργανα τα οποία να κάνουν την ίδια δουλειά και ελπίζω ότι θα το εξετάσει αυτό ο εισηγητή στη συνέχεια. Πάντως χαίρομαι που η Κομισιόν έχει συμφωνήσει να προωθήσει το θέμα αυτό. Αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε επικάλυψη εργασιών. Ε, Πάντω προσβλέπω στην καλή συνεργασία με του άλλου εισηγητέ και με τον εισηγητή. Ο κύριο Χουντή, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν εστερνίζομαι τη θερμή εισήγηση που έκανε ο εισηγητής. Δεν συμφωνώ ότι το θέμα είναι τεχνικό. Το θέμα είναι πολιτικότατο. Επομένως, προκύπτουν δύο κατηγορίες πολιτικών ερωτημάτων και προϋποθέσεων. Πρώτη κατηγορία. Ποιος είναι ο απολογισμός της Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Αν είναι και ας το διευκρινίσει ο εισηγητής τον παρακαλώ διαβάζοντα την έκθεση αν είναι μια επενδυτική τράπεζα που έχει στόχο το κέρδος είναι φανερό ότι με τέτοια νοοτροπία αν κινηθεί και στην περιοχή για την οποία ζητάμε να διευρύνει τις εργασίες πολύ φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρει. Δεύτερο, δεν αποδεικνύεται ότι η οικονομία της αγοράς οι ιδιωτικοποίησεις φέρουν τη δημοκρατία. Μπορώ να σας πω πλήστα όσα παραδείγματα χωρών που έχουν τους κανόνες της δημοκρατίας, της, οικονομικής, της δημοκρατίας της αγοράς, της ε, οικονομία της αγοράς και δεν είναι καθόλου δημοκρατικές. Το αντίστροφο θα έλεγα. Και πολύ φοβάμαι ότι κατά τον απολογισμό της επέδειξε πολιτικές επιλεκτικότητες στο που θα βοηθήσει ή όχι. Τρίτο, αναφέρθηκε και από άλλου συναδέλφους, από τη συναδέλφισσα του Λαϊκού Κόμματος ενδεχομένως, το λέω εγώ με μεγαλύτερη σαφήνεια. Είναι σωστό ότι η τράπεζα με τις δραστηριότητες της έχει εμπλακεί σε έργα που έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα μεταξύ αυτών και προβλήματα στο περιβάλλον. Θα μπορούσα να παριθμίσω μια σειρά ερωτηματικά που είναι της πρώτης κατηγορίας σχετικά τι κάνει αυτή ακριβώς η τράπεζα και αν ο απολογισμός της είναι κάτι το ενθαρρυντικό για να είμαστε, ας το πούμε έτσι, θερμοί για την επέκταση. Και η δεύτερη κατηγορία, με μια σπουδή που δεν την καταλαβαίνω, που δείχνει η Κομισιόν και καλεί και μας να νομοθετήσουμε, ζητάει να επεκταθεί ο ρόλος μιας τέτοιας με πολλά ερωτηματικά τράπεζας σε μια προβληματική περιοχή. Έχουμε κουβεντιάσει προσφάτως με την αφορμή της Αραβικής Άνοιξης πρώτον ότι πρέπει να αλλάξει ο τύπος των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών με αυτές τις χώρες. Διότι εκτός των προβλημάτων των άλλων, ο τρόπος και οι οικονομικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές τις χώρες διήβρυνε τις κοινωνικές ανισότητες. Και ο κόσμος εκεί ξεσηκώθηκε όχι μόνο για αλλά και για το θέμα των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων. Και το δεύτερο, μια τέτοια τράπεζα, αν έχει τα προβλήματα που σας ανέφερα και κινηθεί με το ίδιο στόχο, εύκολα μπορώ λοιπόν να καταλήξω ότι θα είναι ένας ακόμα μοχλός οι προηγούμενες ισχυρές οικονομικές ελίτ των χωρών αυτών μαζί με τη βοήθεια και αυτής της τράπεζας να εκμεταλλευτούν τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους αυτής της περιοχής για την οποία καλείται να διευρυθούν. Αυτά ξέροντας ότι είναι μια πρώτη συζήτηση είναι ορισμένα από τα βασικά ερωτήματα που έχουμε και είμαστε επιφυλακτικοί σχετικά με το τι ακριβώς πρέπει να εισηγηθεί ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι ακριβώς πρέπει να αποφασιστεί. Βεβαίως πρέπει να βοηθηθούν οι χώρες που έχουν προβλήματα, αλλά ανέφερα ορισμένες πλευρές που μας ανησυχούν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Κουλά, εξ της ΑΛΤΕ. Ε, ναι, ευχαριστώ πολύ. Λυπούμε, είχα κάτι άλλο να κάνω. Ω σκιώδη του κειμένου, έχω να πω ότι καταρχήν συμμερίζομαι ε, τα, τα ερωτηματικά κατά πόσο θα πρέπει να διατηρηθούν κάποια θεσμικά όργανα. Είναι καλή αυτή η ερώτηση. Απ' την άλλη μεριά έχω την εντύπωση ότι αν σκεφτούμε του όρου τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων ή της ΕΤΑ, είναι ότι όταν βλέπουμε χώρες που περνάνε από ένα μη δημοκρατικό καθεστώ σε ένα δημοκρατικό θα πρέπει να τις βοηθήσουμε. Και νομίζω ότι με αυτά που γίνονται στη Μεσόγειο θα μπορούσαμε καλύτερα να φανταστούμε τη διεύρυνση της εντολής. Απ' την άλλη μεριά όμως έχω μια ανησυχία όσον αφορά τους όρους και το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογή. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αυτού του τύπου οι διευρύνσεις να είναι σύμφωνες με αυτό το σκεπτικό της βοήθειας στις χώρες που βγαίνουν από μια κατάσταση δημοκρα... ε, δικτατορία. Και ότι τελικά δεν θα πρέπει να καταλήξουμε να έχουμε μια χώρα μη δημοκρατική και να πρέπει να τη βάλουμε επίσης όρις με χώρες που κατέβαλαν κατε... προσπάθησε να το κατεύθυνση αυτή. Ακόμα και στην ε, περιοχή αυτή, ξέρετε τώρα τι λέω, υπάρχουν ε, χώρες που έχουν πάρα πολύ μεγάλο πλούτο ρηκτό, που το παίρνουν οι κυβερνούσες τάξεις και δεν ξέρω γιατί θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει σε κάτι όπου η ίδια η ελίτ της χώρας δεν στρέφεται προς το μέλλον. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε την άγουσα αυτή, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και οπωσδήποτε δεν είναι αυτό μια αυτονόητη ε, λύση. Καταλαβαίνω εκείνος που είναι κάπως πιο επιλεκτική. Αλλά, όπως είπαμε και στην ε, δημιουργία της ε, Ένωση για την Μεσόγειο, ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τη συμβολή μας στις χώρες που καταβάλουν προσπάθειες, ακόμα και αν βέβαια και στις άλλες χώρες βοηθούμε τον τοπικό πληθυσμό και την κοινωνία των πολιτών. Αλλά όταν οι χώρες, οι γειτονικέ Ευρώπης καταβάλουν προσπάθειες προς την κατεύθυνση της δημοκρατίας να μπορούν να βρούν μία υποστήριξη. Είναι καλό αυτό και να δείξουμε και κάποιον ενδιαφέρον για την γειτονίαση με τις χώρες αυτές. Ευχαριστώ κυρία Λούλη. Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη γιατί θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριος Λάμπερς και αυτά που είπε και η κυρία Γκουλάρ. Αυτή η τράπεζα δεν θα πρέπει ποτέ να έχει ε, δημιουργηθεί, αλλά ήταν μια καλή ευκαιρία για τον κύριο Μητερό που ε, ε, έδωσε την πρώτη προεδρία σε ένα φίλο του. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Non, ça c'était euh, surtout euh, dans, dans l'intérêt euh, de la politique αυτό ήταν κυρίως ε, μέσα στα πλαίσια των ε, συμφερόντων πολιτικής ε, προσωπικότητας του κυρίου Μητέρα. Από την άλλη μεριά είπαμε ότι οι δραστηριότητε της ΕΤΑ θα πρέπει να ενσωματωθούν σε κάποιες χώρες και αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό για τους διάφορους λόγους που παρουσιάσαμε ήδη όταν το είχαμε συζητήσει το θέμα προηγουμένως. Ε, εδώ έχουμε δημόσιο χρήμα που σπαταλάται εν μέρη και θα πρέπει να ε, είμαστε συνεπείς με αυτά που λέμε επιτέλους. Δεν πρέπει τη μια φορά να λέμε το ένα και την άλλη φορά να λέμε το άλλο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν έχει πια λόγο ύπαρξης και ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να διαφέρουμε και την εντολή της τράπεζας ΕΤΑ. Α, και η αποστολή θα μπει πού? Δηλαδή, ποιος θα βοηθούσε την αραβική, ε, την αραβική άνοιξη. Μα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αυτό είπαμε. Υιοθετήσαμε μια σχετική τροπολογία που είχα προετοιμάσει και που είχατε και υπογράψει κιόλα. Uh, Κοιτάξτε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Κομισιό να απαντήσει. Κύριε Αστολιάν, μπορείτε να είστε σύνομοι για να δώσω το λόγο μετά στην, ε, στην Κομισιόν. Όταν είχα γίνει αυτές τις πραγματικές για δημιουργία της ήταν πολύ καλή δουλειά, γιατί δημιουργήθηκε ένα μέσο όχι μόνο για, που θα μπορούσε να δώσει πόρους σε κάποια χώρα που βρίσκεται σε ένα μετέχνιο μετάβασης, αλλά για να δοθούν και να δοθεί σωστή υποστήριξη. Είναι πολύ διαφορετική η ΕΤΑ από ότι άλλες τράπεζες, δηλαδή έχει μια τεράστια εμπειρία για την αντιμετώπιση χωρών σε μεταβατική περίοδο όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Λοιπόν, εάν τότε είχαμε σκεφτεί ότι θα μπορούσε η ΤΑ να στηρίξει τις τέων κομμουνιστικές χώρες να μεταβούν στην ε, οικονομία της αγοράς και αν σήμερα θεωρούμε ότι οι αραβικές χώρες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, τότε σαφώς η ΕΤΑ είναι το μέσο που μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις απόψεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Κασόνη. Ε, δημιουργούνται τώρα μια τράπεζα της Αραβικής Άνοιξης. Αυτό το έθιξαν πολλοί όσον αφορά τις επαναλήψεις, ε, ότι κάνουμε τη δουλειά της ε, Διεθνούς Τράπεζας, θίγησαν πολύ σοβαρά θέματα. Ας ακούσουμε λοιπόν την Κομισιόν, παρακαλώ. At the end, if that's okay. Και μετά, κύριε Σιγητά, μπορείτε να επανέλθετε στο τέλος. I, I, I am absolutely open to the conversation with all my colleagues. Είμαι ανοιχτό σε συζήτηση με τους συναδέλφους και αν ε, χρειαστεί να τροποποιήσω κάτι, να αλλάξω κάτι στην έκθεσή μου, είμαι διαθέσιμος, δέχομαι τις ε, προτάσεις, τα σχόλια συναδέλφων. Κύριε Μπίνε, να ζητήσω από την Κομισιόν ε, να μιλήσει προτού να κλείσετε εσείς ε, το θέμα. Κύριος Κασόνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο κύριο Μπίνη αλλά και τους υπόλοιπους αγορητές ε, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που μας προσέφεραν. Θα ήθελα λοιπόν ε, να αδράξω αυτό που είπε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η ΕΤΕ συστάθηκε τη δεκαετία του 1990 για την στήριξη της οικονομίας αγοράς μετά από την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων και αυτή η προσπάθεια στηρίχθηκε από την ΕΤΑ και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ στο ότι εντάχθηκαν και δέκα νέα κράτη, Δυτικά Βαλκάνια και συνεχίζεται ε, με την διεύρυνση προς την Μολδαβία ε, κλπ. Σε ό,τι αφορά την επιτυχία λοιπόν του θεσμού είναι αδιαφεσβήτητο πως ε, πολλά έπραξε προωθώντας μεταρρυθμίσεις ε, για την οικονομία της αγοράς ε, στις χώρες αυτές ε, και συνεχίζει να είναι δραστήρια. Η πρόταση στοχεύει στην τροποποίηση αυτής της συμφωνίας προκειμένου η ΕΤΑ να επεκταθεί στις χώρες της Νοτιού Μεσογείου, κάτι το οποίο στηρίζουν όλα τα κράτη-μέλη και τα 27 αλλά και η διοίκηση της ΕΤΑ. Δέχεται λοιπόν την πρόταση για περαιτέρω διεύρυνση και τώρα υπάρχει διαδικασία κύρωσης από όλα τα μέρη και τους μετόχους και χρειάζεται εδώ να υπάρξει συναπόφαση Συμβουλίου, Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επικύρωση των τροποποίησεων αυτών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμπληρωματικότητα, που ήταν ένα άλλο σημείο που εφήγει από τους ε, αγορητές, θεωρούμε ότι όντω ε, υπάρχει μια συμπληρωματικότητα σε ένα μεγάλο κομμάτι των δραστηριοτήτων ε, της ΕΤΑ. σε τομεί όπου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ιδιαίτερα δραστήρια σε υποδομές κλπ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η άστερη μάλλον εστιάζει ιδιωτικό τομέα, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ. ΕΤΑ είναι μια τράπεζα που βοηθάει στην ε, μετάβαση σε μια άλλη κατάσταση. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρούμε ότι τα είναι ένα στοιχείο κλειδί για τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης. Αλλά και το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του τον Απρίλιο 2011 ε, στήριξε την ε, διεύρυνση προς τον Νότο, διότι η είναι ίσως ε, το εργαλείο μέσω το οποίο αυτά τα κράτη μπορούν να περάσουν σε πιο δημοκρατικό καθεστώτα ε, καθεστώτα που στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Σε ό,τι φορά σημαντικότητα, θα λέγω ότι υπάρχει ένα μνημόνιο κατανόησης ε, τριμερές μεταξύ των δύο τραπεζών και της Κομισιόν. Υπάρχει κλάδι στους οποίους υπάρχει ε, έχουμε συλλογματικότητα και θέλαμε αυτό να επεκταθεί στις ε, αραβικές χώρες όταν επιτευχθούν ε, οι προτινόμενες τροποποίησεις. Τώρα σε ό,τι φορά την διεθνή κοινότητα θα πρέπει να γνωρίζετε πως είναι ιδιαίτερα της είναι ιδιαίτερα προσφυλής μάλλον αυτό η διεύρυνση του, της ΕΤΑ και η διεθνή κοινότητα, όπως γνωρίζετε, θέλει να στηρίξει τις ε, χώρες ε, της Νοτιού Μεσογείου, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και άλλα κράτη προσπαθούν να προωθήσουν το ζήτημα και ελπίζουμε ότι και το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να στηρίξει την πρόταση αυτή. Κύριε Μπίν, θέλετε να προσθέσετε κάτι ή είσαστε ικανοποιημένος. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Νομίζω πως ε, υπόθηκαν όλα. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα έχουμε την παρουσίαση του σχέδιου έκθεση της 20 Μαρτίου. Μετά θα έχουμε προθεσμία για την κατάσταση πολιγίων ε, και θα προχωρήσουμε τον Απρίλιο. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, ευχαριστώ την Κομισιόν. Δίνω το λόγο και πάλι στην Πρόεδρο. disturb the fun. Um, every, every, everybody should know that this is how we... Θα πρέπει να... Ε, σας παρακαλώ. Θα πρέπει να γνωρίζετε πως ε, είναι πολύ ωραίο αυτό το κλίμα που επικρατεί στην Επιτροπή μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σημείο 7, αλλά και στο σημείο 8, διότι θα υπάρξει κοινή συζήτηση. Ελίζα, με ακούς? Ζων Πολ και εσύ. Α, δεν είναι εκτός μικροφώνου ε, κυρία Ελίζα. Ζων Πολ. Θες να ομαδοποιήσουμε τις δύο εκθέσεις ή να εξεταστούν χωριστά μπορούμε να τις ομαδοποιήσουμε. Τις συζητήσουμε ομού και τις δύο, 7 και 8. Το ίδιο μου κάνει. Έτσι κι αλλιώς ε, αποτελούμε συχνά ντουέτο οι δυο μας, ε, συντεύξεις τύπου κλπ. Εντάξει, θα κάνουμε όπως με το six pack. Θα ακούσουμε λοιπόν ε, τους δύο εισηγητές θα περάσουμε στο σημείο 7, ενίσχυση οικονομική και δημοσιονομική εποπτεία των κρατών μελών, τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρέ δυσκολίε αναφορικά με τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ. Ζων Πολ Γκοζέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Το σχέδιο κανονισμού για το οποίο είμαι εισηγητή και που αφορά την οικονομική ενίσχυση των κρατών μελών που γνωρίζουν ή που απειλούνται να ε, με σοβαρές δυσκολίες ε, εντάσσεται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κρίσης και της κρίσης του κρατικού χρέους το οποίο αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να βγάλουμε συμπεράσματα, διδάγματα και να προτείνουμε μια σειρά απολύσεις. Προφανώς ε, τα δύο αυτά ζητήματα το ένα είναι η συγκίτρια Ελίζα, συμπληρώνει το πακέτο για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση που όπως ξέρετε ενεκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο 2011. Ε, πρόκειται το να προσπαθήσουμε να ε, επαναληφθούν σοβαρές κρίσεις οικονομικές που έχουν κοινωνικές επιπτώσεις στις χώρες και μπορούν να έχουν επιπτώσεις και στα υπόλοιπα μέλη της ζώνης ευρώ. Και τα δύο θέματα που μας απασχολούν σήμερα είναι θέματα που αφορούν τις χώρες της ζώνης ευρώ. Το πακέτο των έξι μέτρων θα πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να διασφαλίσουμε την δημοσιονομική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο της ζώνης ευρώ. Αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι σχεδόν ταυτόχρονα με τα δύο κανονισμούς της Κομισιόν, μια διακυβερνητική, διακυβερνητική σύμβαση έχει συσταθεί από τα κράτη-μέλη ευρώ που εγκρίθηκε στο, σε ό,τι το και τώρα θα κυρωθεί από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, στους δύο αυτούς φακέλους. Σε αυτές τις μεγάλες δύο γραμμές λοιπόν η πρόταση της Κομισιόν δεν ε, χρειάζεται, δεν έχει ανάγκη από πολλές ε, επικρίσεις. Θα πρέπει να έχουμε εργαλεία που θα εποπτεύουν καλύτερα τα κράτη-μέλη που ενδεχομένως να γνωρίσουν ε, στο μέλλον δυσκολίες ε, για να τις βοηθήσουν και να τις φέρουν σε μια φυσιολογική κατάσταση τώρα. Απαντώντα ε, απαντώντας στο αίτημα του, κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, το Κοινοβούλιο θέλει τάχιστα να αποφασίσει επί του φακέλου αυτού και να λάβει θέση. Μια που το ομάδα εργασίας του Συμβουλίου ε, μάλιστα τις αρχές του Συμβούλου γνωρίζουμε τα αποτελέσματά της, ε, μπόρεσα να τις λάβω υπόψη μου χωρίς να χρειαστεί να έχουμε μακρές συζητήσεις, χωρίς φυσικά αυτό να απαγορεύει την κατάθεση τροπολογιών από πλευρά σα. Να σας αναφέρω δύο-τρία στοιχεία τα οποία προσανατολίζουν τις προτάσεις μου. Η πρώτη πρόταση είναι να συμπεριλάβουμε στον κανονισμό όλα τα στοιχεία της διακυβερνητικής ε, ε, σύμβασης που μπορεί να ε, προσεγγίσει το σύνολο αυτών των προβλημάτων, των ζητημάτων και να, μην, να χρειάζεται να εξετάσουμε κατά πόσον θα εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό δίκαιο και όχι κάποιο άλλο δίκαιο. Γι' αυτό λοιπόν με την κατάλληλη ορολογία της συνθήκης συμπεριλάβα τα στοιχεία απαραίτητα και μπορώ να σας πω ότι σε αυτή την προσπάθεια έχουμε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα μας βοηθήσει για τις απαραίτητες προσαρμογές. Το δεύτερο στοιχείο της εκθέσεώς μου εισαγάγει την ε, ε, το Συμβούλιο εκεί που δεν ε, είχε συμπεριληφθεί. Αναφέρεται ότι η Κομισιόν μπορεί να πάρει μια σειρά από αποφάσεις ε, χωρίς να συμβουλευτεί το Συμβούλιο. Περίεργος πως το Συμβούλιο δεν έκανε καμία παρατήρηση, ένα σχόλιο επί των σημείων αυτών. Θεωρώ ότι δεν είναι λογικό η Κομισιόν από μόνη της να μπορεί να αποφασίζει δίχως το Συμβούλιο τουλάχιστον να δίνεται να αντιταχθεί. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω μια διαδικασία παρόμοια με αυτή που λάβαμε υπόψη στο πλαίσιο των 6 μέτρων, six pack, δηλαδή το Συμβούλιο να μπορεί να πάρει μια απόφαση με απλή πλειοψηφία και ενδεχομένω να αντιταχθεί, να τροποποιήσει την πρόληψη τη Κομισιόν. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουμε. Τέλο, προτείνω ένα επιπλέον βήμα σε σχέση με τον διδακτικό της ε, Κομισιόν. Και το βλέποντα την κατάσταση στην Ελλάδα παρατηρούμε ότι η χώρα αυτή αντιμετωπίζει μια σχεδόν χρεοκοπία και μια, ένας οίκος αξιολόγησης ε, έλαβε απόφαση περί υποβάθμισης της. Ε, μπορούμε να ε, λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία λέγονται ότι είναι μια έκτακτη κατάσταση. Ποτέ στο μέλλον θα προκύψει μια νέα τέτοια περίπτωση. Εγώ σε ό,τι με αφορά δεν είμαι πεπισμένο ότι αυτό το σκεπτικό είναι βέβαιο. Για το λόγο λοιπόν αυτό προτείνω για την βοήθεια κρατών που ε, ε, ε, εντάχθηκαν σε πρωτόκολλο και έχουν ε, και τη χάνουν μιας να προσθέσουμε λοιπόν ένα επιπλέον βήμα, δηλαδή αυτό τη ε, δημιουργία μια νομική προστασίας των κρατών, που αφού έχουν λάβει ποικίλα μέτρα που, τα οποία του συστάθηκαν, δεν έχουν, κινδυνεύουν να οδηγηθούν στην χρεοκοπία. Αυτό λοιπόν αφορά, μάλλον ε, συνδέεται με το καθεστώς ε, των επιχειρήσεων που ε, αντιμετωπίζουν δυσκολίε όπως και να κάνουμε αυτό που κάνει και μερικοί με το άρθρο 11, δηλαδή τα μέλη της ζώνης ευρώ που βρίσκονται σε μία πληρωμών ή σε πάυση πληρωμών μάλλον που θα οδηγήσει σε μία πάυση πληρωμών, θα πρέπει λοιπόν να μην ε, αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και τις ε, και τις άπειλες που αν τυχόν ε, ε, συμβεί τότε αντιμετωπίζουν κατάσταση ε, χρεοκοπίας. Λοιπόν, να υπάρχουν ε, ρήτρε ε, για ε, default event να παγώνουν και να μην μπορούν να εφαρμόζονται άμεσα. Ζητώ επίσης τα επιτόκια να διατηρηθούν και να μην υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση προς τα άνω των, του κρατικού χρέους και η αξιολόγησης ε, να μην ε, εκδίδουν ε, αποφάσεις και συστάσεις διότι δεν κάνουν τίποτα άλλο στην περίπτωση αυτή από να διατηράσουν τις, τις αγορές. Θεωρώ επίσης ότι είναι χρήσιμο να μπορούμε να εντοπίζουμε τους πιστωτές των χωρών που αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες. Βλέπουμε με την Ελλάδα ότι δεν γνωρίζουμε τους κατόχους των του χρέους της Ελλάδας όπως τα ΣΕΝΤΕΣ ε, ή άλλα, άλλα παράγωγα. Θα πρέπει λοιπόν οι πιστωτές ε, να γίνονται γνωστοί και να γνωρίζουν ε, τι τους περιμένει κατά τον τρόπο. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι αυτές οι διατάξεις αντιβαίνουν του συμβατικού δικαίου αλλά αυτό συμβαίνει όταν ε, αντιμετωπίζουν ε, και στον ιδιωτικό τομέα επιχειρήσεις ε, δυσκολίες. Η δεύτερη ερώτηση με τη σύσταση αυτού του μηχανισμού δεν πιστεύετε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα μπορούν να συμβούν και σε κάποια άλλη χώρα. Απαντώ ναι, αλλά σήμερα η δήλωση ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα δεν μπορεί να συμβεί πουθενά αλλού δεν είναι ε, αξιόπιστο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συμπεριλάβουμε αυτό το εργαλείο προστασίας. Στηρίζομαι πάντως τις ιδέες των ΜΕΝ και το ΔΕ, των μελών της Επιτροπής, για να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα επανόρθωσης ε, του χώρας που αντιμετωπίζει αυτές τις δυσκολίες. Θα πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε να δούμε λοιπόν πώς θα μπορούσαμε να υποχρεώσουμε κάποια κυβέρνηση να λάβει μέτρα στην επεξεργασία των οποίων θα έχει συμμετάσχει και να φροντίσει όλο το σύστημα προστασίας να επιτρέψει στο κράτος ε, να επανορθωθεί σε ένα λογικό χρονικό διάστημα, όχι σε έξι μήνες, σε ένα χρόνο παραπάνω, αλλά αν θέλουμε να προωθήσουμε επενδύσεις θα πρέπει να τις αποφασίσουμε, να τις εφαρμόσουμε και αυτό δεν γίνεται από τη μία, χώρα, από τη μία ώρα στην άλλη. Ευχαριστώ για την ε, μελλοντική συνεισφορά σας. Thank ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προχωρήσουμε τώρα να ακούσουμε την Ελίζα Φερέιρα που είναι η εισηγήτρια για τις ε, κοινέ διατάξεις για την αξιολόγηση των προϋπολογισμών και για τα υπερβολικά ελλείμματα των χωρών στη ζώνη του ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Το κείμενο με το οποίο ασχολούμαι ως εισηγήτρια είναι ο κανονισμός 821 της ε, Επιτροπής. Ένα από τα θετικά στοιχεία της πρότασης ε, είναι ο στόχος του να τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα για τις ε, προϋπολογιστικές διαδικασίες των χωρών μελών. Και θα επιτρέψει στην Επιτροπή να έχει μια καλύτερη επισκόπηση ε, του τι συμβαίνει στην κάθε χώρα και να εντοπίζει ε, σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα και ε, να βρει τρόπο να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι ε, έχω διαπιστώσει να υπάρχει πρόοδος ε, στο κείμενο της ε, Κομισιόν. Θα μπορούσα να αναφέρω κάποια από τα θετικά σημεία. Είμαι ευγνώμων προς τους σκιώδεις εισηγητές για τη συμβολή τους. Ένα θέμα είναι η ανάγκη βελτίωσης του χρονοδιαγράμματος που προτείνεται. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Μιλάμε για το χρόνο που δίδεται στην Κομισιόν για να εξετάσει τα δημοσιονομικά προγράμματα που υποβάλλονται από τα κράτη-μέλη. Υπάρχει και το θέμα του χρόνου που απαιτείται για τον απαραίτητο συντονισμό. Δεν θέλουμε ο συντονισμός αυτός να υπονομεύει την ε, φύση των ε, δημοσιονομικών προγραμμάτων, ούτε τη δυνατότητα των ε, κυβερνήσεων να ελέγχουν τα πράγματα. Ε, αναφέρεται η παράταση της προθεσμίας, ο υποχρεωτικός ε, διάλογος με την Κομισιόν. Αυτά νομίζω ότι είναι χρήσιμα. Δεύτερον, Τα σχέδια ε, δημοσιονομικών προγραμμάτων δεν θα πρέπει να αναλύονται χωρίς να λαμβάνεται η υπόψη η αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εδώ συμπεριλαμβάνονται ε, διάφορες αναλύσεις ε, όπως είναι οι ετήσιες προοπτικές ανάπτυξης, η ανάλυση για τις ε, μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες, καθώς και προτάσεις ε, που έχουν να κάνουν με την απασχόληση. Η όλη ανάλυση λοιπόν θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως ε, ώστε να, μπορούν, ε, ώστε να μπορεί να λαμβάνει υπόψη και τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προς τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενσωματώνουν τις προτάσεις ε, στα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης, στα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλησης, καθώς και στα μεσοπρόθεσμα προγράμματα για την φορολογία. Με βάση αυτή την ανάλυση, Λαμβάνουμε κάθε χρόνο ότι τα σχέδια ε, δημοσιονομικών προγραμμάτων Όλο το πακέτο αυτό ε, θα πρέπει να ταιριάζει. Τα και θα πρέπει να εξετάζεται και στα πλαίσια του ετήσιου προϋπολογισμού καθώς ε, και ε, των πιο μακροπρόθεσμων προγραμμάτων. Θα πρέπει λοιπόν η διαδικασία αυτή να είναι συνεπής όχι μόνο όσον αφορά τον χρόνο αλλά και όσον αφορά τις συστάσεις και προτάσεις που δίδονται. Η επόμενη μου παρατήρηση έχει να κάνει με τη συγκρισιμότητα και το πώς ε, αυτό ταιριάζει στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Στη συνθήκη για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το ε, Fiscal Compact ε, Treaty, υπάρχουν προγράμματα οικονομικής εταιρικής σχέσης, τα οποία θα πρέπει να ενσωματώνουν τις συστάσεις για κάθε κράτος ως μέρος της διαδικασίας για το υπερβολικό έλλειμμα. Αυτές οι συστάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν την συνέπεια με τις μακροοικονομικές ε, συστάσεις ή τις διαθωτικές ε, αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν στο κάθε κράτος μέλος. Τρίτη παρατήρηση. Ε, έχει να κάνει με τον ορισμό των ανεξάρτητων ε, φορέων. Και αυτό είναι κάτι που προκύπτει από την ε, δέσμη των έξι νομοθετικών μέτρων, το λεγόμενο six-pack. Υπάρχουν ε, λοιπόν οικονομικοί φορείς οι οποίοι κάνουν οικονομικές προβλέψεις. Θα πρέπει να είναι απόλυτα διασφαλισμένη η ανεξαρτησία τους καθώς και η αξιοπιστία τους. Αυτό είναι απαραίτητο. Οι προβλέψεις θα πρέπει επίσης να είναι συγκρίσιμες, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να συλλέγει στοιχεία από διάφορες χώρες και από διάφορους φορείς. Καθότι ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις εξουσίες της Κομισιόν, είναι σημαντικό να οριοθετούνται οι εξουσίες αυτές. Είναι πολύ σημαντικό να ε, ε, οριοθετήσουμε τη διαφορά ανάμεσα στην ε, μη συμμόρφωση με τον προϋπολογισμό και ε, σοβαρές περιπτώσεις ε, μη συμμόρφωσης με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν η Κομισιό να δημιουργήσει διάφορες κατηγορίες. Θα πρέπει η Κομισιόν ε, όταν αποφασίζει ότι κάτι δεν συμμορφώνεται να μην είναι αόριστη, διότι αυτό θα οδηγήσει σε αβεβαιότητα. Κάτι το οποίο δεν ε, οδηγεί σε περαιτέρω διαφάνεια, ούτε διευκολύνει την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας. Το πρώτο σχέδιο δημοσιονομικών προγραμμάτων θα πρέπει να ενσωματώνει μια σειρά από πληροφορίες ε, για θέματα δημοσιονομικά. Όχι μόνο αυτό όμως, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και πληροφορίες που να αφορούν τις επενδύσεις την ε, επίτευξη των στόχων για την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς ε, και τις ε, συνέπειες στον προπολογισμό των σχεδίων μεταρρύθμισης, στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Μεταρρύθμισης. Έτσι, ο προϋπολογισμός μπορεί να λαμβάνει υπόψη και διορθώσεις ή τροποποιήσεις που έχουν απαιτηθεί από την εν λόγω χώρα. Θα πρέπει επίσης απαιτείται από το κράτος να ενσωματώσει στο ε, σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος ε, λεπτομέρειες όσον αφορά ε, ένα σχέδιο δημοσίου χρέους. Έτσι μπορούμε να λαμβάνουμε σαφή εικόνα σχετικά με το πώς μία χώρα είναι διατεθειμένη να αντιμετωπίσει πιθανές ανισορροπίες ή ελλείψεις. το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος ε, θα πρέπει να ε, υπόκειται σε κάποιες απαιτήσεις. Ε, δεν θα πρέπει όμως να είναι ανεξάντλητος ο κατάλογος αυτών των κριτηρίων. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία σε συνεργασία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά τον καθορισμό των στοιχείων που θα πρέπει να περιέχει ένα σχέδιο προϋπολογισμού. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε ο κατάλογος αυτός ε, να είναι ανεξάντλητος, διότι μπορεί τελικά να καταλήξουν τα κράτη-μέλη να πρέπει να υποβάλουν τόσες πολλές πληροφορίες που να μην μπορούν να κάνουν την ουσιαστική δουλειά. Τέλος, και αυτό ίσως είναι το πιο ε, σημαντικό μου θέμα, τα κράτη-μέλη απαιτείται να υποβάλουν προς την Κομισιόν ε, και προς την ομάδα του Ευρώ χρονοδιάγραμμα σχετικά με το δημόσιο χρέος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύω ότι πρέπει να καταγράψει αυτά που ε, συμπεριλαμβάνονταν στο ψήφισμα για ε, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Ε, εκεί καταστήσαμε απόλυτα σαφές ότι το σύμφωνο, η δέσμη των έξι νομοθετικών μέτρων, το ΣΥΚΣΠΑΚ δηλαδή, η, η διπλή νομοθετική πρόταση, το ΤΟΥΠΑΚ. Ε, όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε μαζί. Απαιτείται ένας σαφής οδικός χάρτης. αυτά προτάθηκαν στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής το 2011, όπου γινόταν και έκκληση για την άμεση δημιουργία ε, ε, ενός ταμείου αποκατάστασης. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με τρόπο συντονισμένο, ώστε ό,τι κάνουμε εδώ να μην καταστρέφεται από την κερδοσκοπία των αγορών στο δημόσιο χρέος. Είχαμε την ε, δέσμη των, ε, των έξι νομοθετικών μέτρων, τη δέσμη των δύο, το δημοσιονομικό σύμφωνο. Ήρθε λοιπόν η ώρα να πούμε ότι αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή και αποτελούν σαφή δρόμο στον συντονισμό ε, των θεμάτων αυτών και αποτελούν επίσης βήμα προς την άμεση δημιουργία ενός ταμείου αποκατάστασης. Έτσι θα δημιουργήσουμε προστατευτικά τυχή firewall, σε περιπτώσεις ε, υπερβολικού δημοσίου χρέους ε, χωρών ε, της ζώνης του ευρώ. Αυτές είναι οι προτάσεις μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. 14 έχουν ήδη ζητήσει το λόγο, γιατί έχουμε δέκα σκιώδεις για τις δύο εκθέσεις και μετά εκτός από τους σκιώδεις έχουμε τη Σίλβη Λία, και Κούναρ. Και Τιόκο. Άλλος κανείς? Λοιπόν, θα κλείσει εδώ ο κατάλογος των ομιλητών. Πραγματικά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θα παρακαλέσω τους κοιότης να μην μιλήσουν πάνω από τέσσερα λεπτά ο καθένας. Και οι άλλοι ομιλητές ίσως θα έχουν τρία. και μετά τέσσερις ε, κάθε ένας από τους ηγητές στο τέλος. Παρακαλώ τηρήστε το χρόνο αυτό για να μην έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, δεν θα εξετάσουμε τώρα με τη σειρά των ομάδων, αλλά για την κάθε έκθεση πάλι και δύο εκθέσεις ταυτόχρονα του τους δύο σχεδόν. Για την έκθεση Πολ Ελίζα, εσύ είσαι νομίζω η πρώτη σκιώδης, άρα τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ, Σέραν. Αυτή η έκθεση του Ζωοπόλ Γκοζές είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. λέει ότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτή η προστασία κεφαλαίου 11 που έχουν στη ΣΥΠΑ για να μπορούν να προστατεύουν οι χώρες και νομίζω ότι αυτό πράγματι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η ιδέα έχει ιδιαίτερη σημασία. Ταυτόχρονα όμως θεωρώ ότι ίσως υπάρχουν κάποιες δυνατότητες βελτίωσης της πρότασης. Ε, γενικά όμως η ιδέα του μου φαίνεται πάρα πολύ θετικός. Θα ήθελα να φέρω τέσσερα στοιχεία όπου κατά τη γνώμη μου μπορούν να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις. Πρώτο, πρόκειται για ένα σκληρό σύστημα για εκείνες τις χώρες που έχουν πραγματικές δυσκολίες. Απ' την άλλη μεριά όμως νομίζω ότι δεν είναι πολύ ξεκάθαρο το τι εννοούμε όταν λέμε δυσκολίες. Ο συνάδελφος Κοζές ανέφερε στο 7α και στο 7γ κάποιους λόγους. Αλλά, εάν κοιτάξει κανένα το διατακτικό, πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει και κάτι άλλο, δηλαδή να φέρτε, παραδείγματος χάρη μια σταδιακή επιδείνωση της κατάστασης ή θα πρέπει να υπάρχει κάποια διαδικασία σταδιακή, σταδιακή πριν ε, μια χώρα να περάσει στο καθεστώς της Τρόικα αν θέλετε και αυτό το στοιχείο εκκίνησης μέχρι να περάσει κανένα αυτή την εποπτεία θα πρέπει σιγά σιγά να οριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια, ούτως ώστε ο καθένας να καταλαβαίνει πότε περνάει κάποια χώρα σε εποπτεία. Και για να αποφύγουμε να υπάρχουν πάρα πολύ μακρά όρια διακριτικής ευχέρειας. Δεύτερη σκέψη. Υπάρχει και κάτι καινούριο σε αυτό το κείμενο όσον αφορά τους όρους για τις ε, αιτήσει ενίσχυσης από κάποιες χώρες. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Μία χώρα μπορεί ενδεχομένω να υποχρεωθεί, για να το πω έτσι, να ζητήσει βοήθεια από κάποια από τα κοινοτικά ταμεία. Αυτό όμως δεν συνοδεύεται από όρους βάσει των οποίων θα πρέπει να υπάρχει μια θετική απάντηση του Ταμείου. Δηλαδή μια χώρα θα υποχρεωθεί να υποβάλει μια αίτηση και πού είναι το αντίβαρο. Δεν μου φαίνεται αυτό σωστό. Ίσως θα έπρεπε να είναι μια προσφορά προς μια χώρα να τύχει βοήθειας. Ας πούμε, άμα ζητήσει βοήθεια, ναι, ναι, ε, να μην τη συνεννηθούμε. Και τελειώνω, πρόεδρε. Ε, κεφάλαιο 11. Ε, μας λείπουν νομίζω κάποιες λεπτομέρειες και υπάρχει κάτι που δεν κατάλαβα καθόλου γιατί λέγεται ότι οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους και όχι το κράτος μέλος θα πρέπει να κληθεί να υποβάλει τις πληροφορίες. Στο κεφάλαιο 10 θα πρέπει να δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις. Εκτός από τις λεπτομέρειες αυτές όμως το κείμενο είναι πάρα πολύ καλό. Με συγχωρείτε, 45 δευτερόλεπτα μακρηγόρησα. Ωραία. Μάριον Τάισεν. Δεν είναι εδώ. Μιλάει κάποιος εξ ονόματος της Μαρίαν. Όχι. Ωραία. Όχι, ε, ναι, η Μανιτά δεν είναι παρούσα γι' αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια για την έκθεση της Ελίζας. Θα υποβάλει ε, αν δεν το έχει κάνει, ποιε είναι οι διατάξει ε, που δεν είναι οι κατάλληλε κατά τη γνώμη του. Αλλά εντάξει, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Άλντε. Άγγλων και μετά Ρήμον Τρεμόζα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Είμαι ισχυώδης για την έκθεση του κυρίου Γκοσέ και θα μπορέσω να είμαι κατά δυνατόν σύντομο. Καταρχήν, όσον αφορά την ιδέα του Ζαν Πολ να συμπεριληφθούν στοιχεία της ε, συνθήκης των διεθνών συμφωνιών. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Η ομάδα μας είναι υπέρ αυτή τη προσέγγιση που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ θετική. Αυτό είναι γενικό σχόλιο. Υπάρχουν μετά κάποια θέματα που θα πρέπει να αναλυθούν εις βάρος Καταρχήν, γενικά η Κομισιόν στην πρότασή της χορηγεί περισσότερες εξουσίες σε αυτόν. Αυτό είναι κάπως πολύ λεπτό. Το μάθαμε όταν διαπραγματευτήκαμε ε, το Six Pack, ότι αυτό πρέπει να είναι πολύ λεπτό, ιδίω όσον αφορά την πλευρά του Συμβουλίου. Από την άλλη μεριά ξέρουμε ότι οι χώρες να αλληλοελέγχονται δεν είναι πολύ θετική επίσης λύση. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί από την άλλη μεριά με τις προτάσεις που δίνουν στην Κομισιόν τις αρμοδιότητες αυτές και τις εξουσίες αυτές. Γιατί τελικά η χώρα που είναι το αντικείμενο της ε, αυξημένης ε, εποπτείας ε, θα πρέπει να δει πώς θα το αντιμετωπίσει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω περισσότερα, θα πρέπει να το σχολιάσουμε κάποια στιγμή πιο αναλυτικά ιδίως όσον αφορά την ατμόσφαιρα που διέπει το Συμβούλιο. Ένα άλλο θέμα που αφορά τη συνθήκη μέσω της Διεθνούς Συμφωνίας είναι η διεθνής, είναι αιτήσια, συγγνώμη, ισορροπία που επιτρέπει το 0,5 διαθετικό έλλειμμα στο κράτος μέλος. Δεν ξέρω κατά πώς θα πρέπει να το πούμε έτσι ή όχι γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό 0,5% είναι κάτι που έχει ήδη προσαρμοστεί στην οικονομική κατάσταση. Το θέμα είναι λοιπόν, θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι παρόλο στους προσωμαγές της κατάστασης επιτρέπουμε στις χώρες να έχουν διαστατικό έλλειμμα. 0,5 είναι μικρό. Δεν βοηθάει και πάρα πολύ δηλαδή. Και γι' αυτό δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το 0,5% πρέπει να το κρατήσουμε. Εάν λοιπόν θέλει κανένας να είναι ευθυγραμμισμένος με την συνθήκη, το 0,5% είναι σωστό. Εγώ δεν συμφωνώ παρόλο που πρόκειται από τη συνθήκη. Ένα σύντομο σχόλιο όσον αφορά τα διευθυντικά ταμεία και την διακοπή των πληρωμών. Ξέρουμε ότι είναι πολύ επίκαιρο το θέμα αυτό, αν δούμε τι γίνεται στην Ουγγαρία. Το συζητήκαμε διαμακρών στις διαπραγματεύσεις για το Six Pack ε, όταν εξετάστηκε η δική μου έκθεση και δεν υπήρχε τότε πλειοψηφία. Τώρα όμως νομίζω θα πρέπει να ανοίξουμε λιγάκι τη συζήτηση. Γιατί ίσω υπάρχουν αιτιολογήσεις, είναι πολύ λεπτό το θέμα, το καταλαβαίνω αυτό, το ξέρω. Η Επιτροπή των Περιφερειών μας έστειλε ένα πολύ κριτικό email για το θέμα αυτό σήμερα. Τέλο, όσον αφορά τι δύο πρωτοβουλίε, θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Η Ελίζα είπε ότι είναι θετική υπέρ. Εγώ δεν έχω διαφωνίε αρχή, αλλά αναρωτιέμαι τι σημαίνει και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Έχω κάποιες ε, αμφιβολίες. Ε, πρέπει να το συζητήσουμε λοιπόν διαμακρον Αυτά τα τέσσερα λεπτά έληξαν. Ευχαριστώ. Προς ευχαριστώ Ευχαριστώ Σάρων. Είμαι σκιώδης ε, στην έκθεση Φέιρα. Νομίζω ότι αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για να θέσουμε στο επίκεντρο μια ιδέα που θα ήθελα να υποβάλω. Μιλάω για την πρόταση δημιουργίας ενός ε, ταμείου διάσωσης, ε, Redemption Fund. Είναι γερμανική ιδέα αυτή. Κάτι το οποίο θα απορροφά όλο το χρέος άνω του 60%. Το ταμείο αυτό θα έχει ε, ένα χρονικό ορίζοντα 20-25 ετών και δεν απαιτεί αλλαγές στι συνθήκε. Αυτό το Ταμείο θα επιτρέψει τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ε, σοβαρό κίνδυνο να χρηματοδοτεί το χρέος και να μπορέσει να χορηγεί ως εκ τούτου κονδύλια για ανάπτυξη. Καλωσορίζω το αυτό που είπε η κυρία Φεραίρα για το θέμα της Δημοσιονομική Πειθαρχία και νομίζω ότι μπορούμε να πείσουμε τον κύριο Γκοζές και το ΕΛΚ έτσι ώστε να εστερνιστούν αυτή την θέση. Πιστεύω ότι το ελληνικό χρέος ε, πόρο απέχει από το να έχει διευθετηθεί και θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι πραγματικά προχωράμε με εγωργό βηματισμό για μια οικονομική και δημοσιονομική ολοκλήρωση. Τα ευρωμόλογα δεν αφορούν τη σημερινή κρίση, θα αφορούν την μελλοντική, την επόμενη και κατανοώ τον προβληματισμό των ε, κράτων μελών. Είμαι από την Ισπανία, μια χώρα που δεν μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι μια χώρα που που εφαρμόζει μια καλή πρακτική. Είχαμε τα, τα αποτελέσματα του περσινού ελλείμματος 8,5% αντί το 6%. με τόση πόρα έχουμε ακόμα από τα Eurobonds, από τα ευρωομόλογα. Αναφέρω ότι τα προτινόμενα στις ε, δύο εκθέσεις ε, είναι πάνε προς την κατεύθυνση. Και μια προσωπική άποψη θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει το ρόλο της Κομισιόν σε αυτό το πακέτο. Κατ' εμέ, ο μόνος τρόπος για να επιβάλλουμε κανόνες είναι να διασφαλίσουμε πως τα κράτη-μέλη δεν είναι αυτά που μόνα τη αποφασίζουν η Κομισιόν, είναι ο μοναδικός πρωταγωνιστής ανεξάρτητος και που ενεργεί με βάση αντικειμενικά πρότυπα. Αυτή είναι η άποψή μου προσωπική. Θα πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να έχει τον τελευταίο λόγο για επιβολή κυρώσεων αναφορικά με το υπερβολικό έλλειμμα των κρατών μελών. Θα πρέπει να διαδραματίσει έναν υποπτικό ρόλο για να διασφαλίσει την ουδετερότητα και την αντικειμενικότητα σε όλες, ε, και την αναλογικότητα όλων των κυρώσεων. Τέλος, ε, και συμφωνώ με την τροπολογία σας 21 Ορισμένε έκτακτε καταστάσει θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη προκειμένου να αξιολογήσουν τη συμμόρφωση με τα προγράμματα συμμόρφωση ε, και, και προσαρμογή. Ε, συμφωνώ επίση να αποκτήσει μεγαλύτερο ρόλο του Κοινοβουλίου σε ό,τι φορά την δημοκρατική λογοδοσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην ομάδα ECR και έχει το λόγο 8 λεπτά γιατί θα μιλήσει για δύο εκθέσεις. Καλωσορίζω γενικά τη πρωτοβουλία τη Κομισιόν για την οικονομική διακυβέρνηση, αλλά φτάνουν με 10 χρόνια καθυστέρηση. Ε, όλα αυτά που τα οποία προτείνονται είναι προπόθεση, ε, αλλά είμαι συγκρατημένα αισιόδοξο. Ε, η Γερμανία τώρα έχει καταστεί το το ισχυρότερο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, μετά τις μεταρρυθμίσεις που έκανε σε πολλά θέματα, ακόμη και στην αγορά εργασίας. Έχουμε το παράδειγμα επίση του Μάριο Μόντι και του Μαριάνο Ραχώη στην Ισπανία, οι οποίοι έχουν δεσμευθεί να προωθήσουν ε, μεταρρυθμίσει. Η ε, μεγαλύτερη απειλή μπορεί να προέρχεται από τη Γαλλία. Ο υποψήφιος πρόεδρος Φρανσουάν Ολάντ είπε ότι θα ε, αναδιαπραγματευτεί το Δημοσιονομικό Σύμφωνο αν εκλεγεί. Ε, σήμερα διάβασα στο ίντερνετ ότι θα αυξήσει στο 75% την, την φορολογία για ε, τους ανθρώπους με υψηλό εισόδημα. Όταν αυξήθηκε το όριο στο από το 60 στα 62, ο jean Λουκ Μελανζόν, ο ηγέτης ε, της Front de θεώρησε ότι αυτό είναι το τέλος ε, του γαλλικού τρόπου ζωής. Είναι συνάδελφος από ό,τι φαίνεται ο κ. Μελανζόν, αλλά εγώ δεν τον έχω τίποτε. Στις ε, προσεχείς ε, προεδρικές εκλογές ε, λοιπόν διακυβεύεται και το ευρώ και ο γαλλικός τρόπος ζωής. Ε, όσον αφορά την έκθεση του κυρίου Γκοζές, ε, προτείνει να ε, τεθεί υπονομική προστασία ένα κράτος μέλος εάν κινδυνεύει να χρεοκοπήσει. Τέτοιες προτάσεις έκανε η Ολλανδική κυβέρνηση πέρσι. Εγώ καταλαβαίνω τη λογική και θα ήθελα να προσθέσω ότι αν ένα κράτος μέλος δεν θέλει να χωρίσει την κυριαρχία του, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει από την ζώνη του ευρώ. Και ρητή αναφορά στη δυνατότητα αυτή θα ε, ε, ήταν κάτι που επικροτούμε. Και επίσης ε, όσον αφορά το καθεστώς προστασίας για τα χρεωμένα κράτη, Εμένα μου κάνει εντύπωση η πρόταση του κυρίου Γκοζέσε να περιορίζεται η πρόσβαση στα διαφορετικά ταμεία. Συμφωνώ ότι θα πρέπει η πρόσβαση των αμαρτωλών να εξαρτιέται από προϋποθέσεις αλλά ε, ε, αραιώνεται πολύ η ε, πρότασή της Κομισιόν από την κυρία, Κομισιόν, από την κυρία ε, από την κυρία Φερέιρα. Ο κύριο ε, Γκοζέ προσπαθεί να σφίξει τα μέτρα, ενώ η κυρία Φερέιρα τα αποδυναμώνει επιπλέον. Η Κομισιόν μπορεί να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να αλλάξουν τα σχέδια ε, προπολογισμού του μόνο εάν δεν καλύπτονται επαρκώ οι συστάσει. εγώ βλέπω να υπάρχει ε, κίνδυνο να υπονομεύσουμε το στόχο του προτινούμενου κανονισμού. Η κυρία Φερέιρα, σε περίπτωση ε, οικονομική κάμψη, προτείνει ε, προσαρμογή του κανόνα για το χρέος και η τελευταία μου παρατήρηση ε, έχει να κάνει με ένα θέμα στο οποίο θέλει να επιμείνει η ομάδα μου. Μπορείτε να ε, μιλάτε λίγο πιο αργά. Ναι, προσπαθούσα να ολοκληρώσω μέσα σε τέσσερα λεπτά. Η κυρία Φερέιρα θέλει να να εισάγει την, ε, την εποπτεία του προϋπολογισμού, ε, ε, αλλά αυτά όλα αποτελούν ηρωνία. Το να επιδοτούμε κράτη-μέλη με υψηλό χρέος υπονομεύει τη ζώνη του ευρώ και δεν έχει διαφορά αν ε, ονομάσουμε την πολιτική αυτή ομόλογα σταθερότητας. Κάθε χώρα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες ε, μιας νομισματικής ένωσης σεβόμενη την ε, αρχή περί μη διάσωσης καθώς και τους κανόνες καλή οικονομική διακυβέρνησης. Αν δεν τα προσέξουμε όλα αυτά θα διαβρωθεί το νόμισμά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα προχωρήσουμε τώρα στους σκιώδεις εισηγητές των Πρασίνων. Παρακαλώ. Um, Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το σχέδιο έκθεσης, ε, καταρχήν ε, για την πρόταση, ε, πάνω στην πρόταση της Κομισιόν και κατόπιν στο σχέδιο έκθεσης του jean Πολ Gauzès. Η έκθεση αυτή μπορεί να είναι προς το παρόν η τελευταία ε, ευκαιρία στα πλαίσια της κρίσης ε, να ε, έχουμε λίγη δημοκρατία, διότι με, το, με την δέσμη των έξι νομοθετικών μέτρων εισάγαμε κάποια μέτρα, έχουμε κάποιες υποχρεώσεις λογοδοσίας, αλλά δημοκρατικό έλεγχο δεν έχουμε υπό τη μορφή αυτή και γι' αυτό η έκθεση αυτή αποτελεί ευκαιρία να θέσουμε ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να είναι απαραίτητο εάν δει κανείς ε, πώς έχει η κατάσταση στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και στην Ιταλία. Ε, αν δει κανεί δηλαδή πώ έχει εξελιχθεί η κοινωνική κατάσταση στι χώρε αυτέ, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τα, τα προγράμματα αυτά επιτυχία. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει κοινοβουλευτικό έλεγχο. Για μένα τίθεται όμω και το ερώτημα εάν ε, το πεδίο εφαρμογή αυτού του κανονισμού ε, έχει επιλεγεί σωστά. Εάν μόνο τα κράτη-μέλη του ευρώ είναι αυτά όπου χρειαζόμαστε αυτόν τον ενισχυμένο δημοκρατικό έλεγχο. Μήπως ε, χρειαζόμαστε να εξετάσουμε και πιο προσεκτικά τι γίνεται με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες όπως είναι η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Λετωνία. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να το κοιτάξουμε αυτό. Τίθεται και το θέμα του νομικού πλαισίου αλλά ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν πώς έχει καταλήξει σε αυτόν τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάζουμε και τις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ. Ε, η Μεγάλη Βρετανία δεν βρίσκεται στη ζώνη του ευρώ, πάλι δεν λαμβάνει ε, τέτοιες επιδοτήσεις, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος και όσον αφορά αυτά που γίνονται στην Ανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, όσον αφορά το θέμα ποιο θα πρέπει να εμπίπτει στο πλαίσιο, πιστεύουμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο, κανένα όμω δεν θα πρέπει να αποφασίζει μόνο του. Πιστεύω ότι η ιδέα να έχουμε αντίστροφη ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο είναι ο σωστό ε, μηχανισμός λήψης αποφάσεων. Ε, συμφωνούμε δηλαδή εδώ με τον Τζον Πολ Γκοζές. Το δεύτερο θέμα είναι ότι ε, έχουμε την συμμετοχή διαφόρων ε, θεσμικών οργάνων όπως είναι της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όχι όμως των εποπτικών αρχών που έχουμε δημιουργήσει μαζί. Στο άρθρο 3 είναι απαραίτητο να συμπεριλάβουμε και τις άλλες εποπτικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας των Τραπεζών. Θα πρέπει εδώ να συμμετέχουν όλες οι εθνικές εποπτικές αρχές και η ΕΙΟΠΑ διότι η οικονομική ε, κρίση ε, έχει ε, εισβάλλει και στον τομέα των ασφαλίσεων. Και όσον αφορά το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, οι στόχοι των στρατηγικών απασχόλησης και ανάπτυξης θα πρέπει να ενσωματωθούν. Και παράλληλα με το πρόγραμμα χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά το είδος τεχνικής υποστήριξης που θα πρέπει να παρέχεται. Και εδώ μας ενδιαφέρει και η καλή διακυβέρνηση, η λειτουργία του κράτους, ε, καθώς ε, και ε, φορολογικές διοικήσεις που να λειτουργούν καλά. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αναφέρουμε ρητά. Βρίσκουμε σωστό το Ευρωπαϊκό ε, Εξάμεινο και το πρόγραμμα για την εξάλληψη των ε, ανισορροπιών ε, να συνδυαστούν ώστε να μην έχουμε επικάλυψη των εργασιών. Είναι καλό αυτό που έχει αποφασίσει η Κομισιόν. Όσον αφορά όμως τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, το κεφάλαιο 8 δηλαδή, στον τομέα αυτών δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις χώρες, διότι δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε κάποιες χώρες, διότι θα έχουμε πίνακες τις χώρες που έχουν κρίση, το οποίο δεν έχει κανένα νόημα. Ε, επίσης, ε, όλες οι εκθέσεις, ιδιαίτερα οι τριμηνιές, ε, στο, κεφάλαιο, στο άρθρο 6.3 καθώς ε, και οι εκθέσεις ε, σχετικά με την επιστοληπτική ικανότητα στο άρθρο 5 πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δημοσιεύονται. Ε, δεν, μπορούν, δεν μπορούμε να τα λαμβάνουμε αυτά από τους Financial Times ή από αλλού. Εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουμε τα στοιχεία αυτά και... Κατά την εκπόνηση των εκθέσεων αυτών πιστεύουμε θα πρέπει να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών οτι και η κοινωνική εταίρη. Τέλος, επικροτούμε την πρόταση του Ζαν Πολ σύμφωνα με το άρθρο 11 το κεφα... Ε, να προβλέπουμε έναν ε, μηχανισμό παρόμοιο με αυτόν στο κεφάλαιο 11 που έχουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ευχαριστώ. Ήδη ξεπεράσει το χρόνο σας κατά 1,5 ε, λεπτό. Φιλίπ, μπορείς να εξηλεωθεί εσύ για τους πράσινους. Πέντε παρατηρήσεις για την έκθεση Φερέιρα. Πρώτον, Θέλουμε να έχουμε ισορροπία μεταξύ οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη και ανάπτυξη και ε, βιωσιμότητα. Αλλά ε, είδαμε ότι υπάρχουν ε, οι ρήτρε ε, μόντι, γιατί πρέπει όμω να επαναλάβουμε κάτι τέτοιο, διότι θέλουμε ότι η Κομισιόν να μην το αγνοεί όπω το πράττει τώρα στην Ελλάδα μα ε, το να περι, μισθών, αυτό δεν είναι θέμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά του κοινωνικού εταίρου. Και αυτό αναφέρεται ρητά στι συνθήκε. Να επιθυμεί η Κομισιόν λοιπόν ότι θα πρέπει να ενεργεί μέσα σε συγκεκριμένα όρια. Και όχι ανεξέλεγκτα. Όπω είπε και ο Σβέν, στρατηγική 2020, η στρατηγική ανάπτυξη ε, και απασχόληση έχουμε, χρειάζεται να έχουμε προπολογισμού στου οποίου καταρτίζουν τα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να βλέπουμε σαφώ τον σχέση μεταξύ αυτών των προπολογισμών και τη στρατηγική 2020. Τρίτον, πρέπει να ενισχύσουμε την δημοκρατική πτυχή. Και αυτό σημαίνει αλλαγέ στο χρονοδιάγραμμα, διότι όσο έχει το χρονοδιάγραμμα τα Εθνικά Κοινοβούλια αποφασίζουν για προπλογισμού, ε, αλλά δεν πρόκειται για μια ουσιαστική δημοκρατία, διότι τα Εθνικά δημοκρατία, ε, Κοινοβούλια παίρνουν αυτά τα προπλογισμού που έχει συντάξει η Κομισιόν και το ΚΡΑΡ και η κυβέρνηση και του λένε ή το δέχεστε ή το απορρίπτεται. Αυτή δεν είναι δημοκρατία ευρωπαϊκή. Είναι του Παϊκίνου, όχι των Βρυξελών. Τώρα συζήτηση με τους ε, κοινωνικούς εταίρου και με συμμετοχή αυτών. Τελευταίο σημείο πιστεύουμε ότι η Κομισιόν χρειάζεται να καταρτήσει μεθόδους και μοντέλα δημόσια. Μα αυτό θα μου πείτε δεν είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό διότι πριν από δύο χρόνια η Κομισιόν ήταν κα... Ε, δεν ε, έκρινε ότι η Ελλάδα είχε καταλήξει σε μια αδυναμία, θα καταλήξει σε μια αδυναμία πληρωμών. Και όμως έτσι είχαν τα πράγματα και το ξέρουμε, διότι έτσι εκθέτουμε τους ε, Ευρωπαίους πολίτες σε τεράστια έξοδα. Χρειαζόμαστε λοιπόν απόλυτη διαφάνεια και σε επίπεδο κομισιών. Και θα κλείσω εδώ λέγοντας ότι Λέτε πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη εξουσία στην Κομισιόν. Λέω, δημοκρατία σημαίνει ε, εκλογές, ε, έλεγχη και ισορροπίες. Σε οποιοδήποτε πολιτικό σύστημα δώσετε ανεξέλεγκτη εξουσία. Δεν βρισκόσαστε πλέον σε δημοκρατία. Μπορεί να σας αρέσει αυτό που κάνει η Κομισιόν, μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά όπως και να έχει το ζήτημα, χρειάζεται να έχουμε ελέγχους ε, και ισορροπίες. Δεν μπορεί η Κομισιόν να δρά ανεξέλεγκτα, διότι αυτό δεν οδηγεί στη δημοκρατία. Εμείς ως βουλευτές πρέπει να φροντίσουμε να, το, να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Εμείς ε, δεν θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι που θα πούμε γεια, σου, γεια στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Ωραία. Περνάμε τώρα στην ΚΟΕ. Ο κ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αναφέρομαι στην εισήγηση, στην έκθεση του αγαπητού συναδέλφου Γκοζές. Θα είμαι σύντομος. Τι μας καλεί η έκθεση. Μας καλεί να παρακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον παροξισμό της Ευρωπαϊκής της Κομισιόν που με αλλεπάλληλα αντικοινωνικά νομοθετήματα τα οποία ορισμένα επικαλύπτουν τα υπόλοιπα σε ένα συνεχή αγώνα. Το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης έκανε πιο αυστηρό το σύμφωνο σταθερότητας. Και τώρα το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης συν οι δύο κανονισμοί, η έκθεση των οποίων καλύπτει, η εκθέση των οποίων καλύπτουν οι συνάδελφοι, θέλουν να κάνουν πιο αυστηρό το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης. Η άποψή μας είναι ότι είναι λάθος κατεύθυνση, λάθος συνταγή και δεύτερο σημείο ο συνάδελφος του οποίου εκτιμώ τη σοβαρότητα, μπορεί να μην συμφωνώ, διαπιστώνει και αντιφάσεις και ουσιαστικά υπογράμισε ότι μέσα στην έκθεσή μας πρέπει να περιλάβουμε και το νέο σύμφωνο, το δημοσιονομικό σύμφωνο, το οποίο είναι εν εξελίξη αν υιοθετηθεί. Σήμερα, συνάδελφοι, από ό,τι άκουσα, η Ιρλανδία θα κάνει δημοψήφισμα για αυτό το θέμα, αλλά πρέπει κάπου να συμβιβαστούν αυτά. Άρα αυτό που επικαλύπτεται κάπου που πρέπει να βρεθούμε σε κοινό σημείο είναι ορισμένες από τις αντιφάσεις. Το αποτέλεσμα είναι πολιτικές καταστροφικές. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα ε, ε, δεν ερμηνεύεται καλά ενδεχομένως, αλλά εδώ έχουμε φαινόμενα ύφεση σχεδόν σε όλη την Ευρωζώνη. Η οίκη πιστοληπτικής ικανότητας ε, ε αξιολόγησης δεν υποβαθμίζουν μόνο την Ελλάδα, έχουν υποβαθμίσει τουλάχιστον ορισμένοι από δάφτου, ορισμένε από τι άλλε χώρε, και επομένω η κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Τώρα θα αναφερθώ σε δύο-τρία σημεία αυτή καθ' αυτή τη έκθεση, γιατί την ε, πρόσεξα έτσι πιο σοβαρά. Πρώτον, μου έκανε εντύπωση γιατί ο εισηγητής στην τροπολογία 1 βγάζει την αναφορά εκτός, εκτός του πλαισίου της Ένωσης. Δηλαδή ζήτησαν οι χώρες χρηματοδοτική υποστήριξη εκτός του πλαισίου της Ένωσης. Εδώ τα ερωτήματα στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται καθώς στην έκθεσή του αποδέχεται και δεν ξέρω ποιος τα αποφάσισε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν αυτό είναι το εκτός του πλαισίου της Ένωσης, είναι θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω αναφερθεί αρκετές φορές σε αυτό το θέμα, δεν έχει δοθεί απάντηση, το θίγω μόνο από την άποψη. Αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι θεσμός της Ένωσης, ας το πούμε ποιος το αποφάσισε. Αν δεν είναι θεσμός και επομένως η συνεργασία μαζί του είναι διεθνή συμφωνία, πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποια στιγμή, σύμφωνα με το άρθρο 218, εμείς, παράγραφος 6, να μιλήσουμε. Το δεύτερο που θέλω να πω, αν κατάλαβα καλά, ο σοβαρός, ξαναλέω και με ε, εισηγητής μας, καταλαβαίνει τις ακρότητες της του σχεδίου κανονισμού της Κομισιόν και αν είναι σωστή μετάφραση και συμφωνώ βεβαίως όσον αφορά στην τροπολογία 3 λέει να διαγραφεί τούτο εδώ το πράγμα. Αν ο εισηγητής μας το εισηγείται, δηλαδή ότι δεν πρέπει να στερούνται αυτές οι χώρες που έχουν προβλήματα από τα διαρθρωτικά ταμεία και είναι αυτή η άποψή του, συμφωνώ, είναι μια αγριότητα. Δεν θα βγάλει άκρη, αν είναι έτσι. Αν είναι το αντίθετο, δεν συμφωνώ με όποιον εισάγει τέτοιε εισηγήσει. Εν πάση περιπτώσει, η εποπτεία με αυτά και με αυτά γίνεται ενισχυμένη, γίνεται προληπτική και γίνεται και αιωνία. Και επομένως δεν θα λύσει το πρόβλημα. Τελείωσα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Thank you. Εγώ σας ευχαριστώ. Τέσσερα λεπτά ακριβώς. Πολύ καλά. Μικουέλ. Νομίζω θα καταφέρω να τελειώσω σε ένα λεπτό. Έχω τρεις παρατηρήσεις όσον αφορά την έκθεση της κυρίας Φερέρα, καταρχήν. Η έκθεση Κοζές και Φερέρα είναι μία δέσμη ε, κοινή, αν θέλετε. Το πρόβλημα που έχω με την έκθεση της Ελίζα είναι ότι αντιμετωπίζει θέματα που ίσως δεν θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν από κοινού. Μετά, το χρονοδιάγραμμα. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα ουσίας. Έχουμε την ιδέα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τώρα θέλουμε να υπάρχει μια διαδικασία ελέγχου αλλά όχι ανά αλλά ανά έτος, όπως παραδείγμα και δημοσιονομική διαδικασία. Και αυτό οδηγεί σε ένα δημοκρατικό πρόβλημα ουσίας. Έχουμε μια κυβέρνηση που το Σεπτέμβριο υποβάλλει κάποιες ε, δημοσιονομικές προτάσεις βάσει ενός ευρωπαϊκού ε, προσανατολισμού συγγνώμη, και μάλιστα ε, κατόπιν μιας ευρωπαϊκής συζήτησης για τις δημοσιονομικές προτεραιότητες ανακράτως. Ένα αυτό. Άλλο αυτό όμως που θέλουμε σήμερα. Να εισαγάγουμε μεταξύ της στιγμής κατά την οποία η κυβέρνηση υποβάλλει την πρόταση για τον προπολογισμό και τη στιγμή κατά την οποία πρόκειται να ψηφιστεί στο, στη Βουλή έχει μια καινούρια διαδικασία προσθεθεί που ίσως οδηγήσει το κράτος στο να επανεξετάσει την θέση του. Άρα το ε, Εθνικό Κοινοβούλιο είναι μια αίθουσα απόϊχου των Βρυξελών ίσως. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία. Ακόμα και σε μια ομοσπονδιακή χώρα, ένα παραπάνω μέσα σε μια ε, ενότητα όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, που θα ήθελα να αναφέρω. Συμφωνώ. Πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός και ε, συντονισμός των στοιχείων για τα χρέη και να πούμε ότι το ποσό εκκίνησης δεν επιτρέπεται να είναι ίσο με το σφαιρικό ποσό για τα ευρωομόλογα. Και αυτός ο μηχανισμός ε, φορολόγησης που μειώνει τη δημοκρατία σε εθνικό επίπεδο και αφαιρεί από τα εθνικά κοινοβούλια το πιο σημαντικό τμήμα της ε, εξουσίας τους για αποφάσεις δηλαδή τη δημοσιονομική εξουσία. Πρέπει λοιπόν κατά τη γνώμη μου αυτή η λογική ε, που καταπνίγει τη δημοκρατία θα πρέπει να μην ακολουθεί. Δηλαδή υπάρχουν πολιτικές διάσωσεις που είναι τελικά καταστροφή για τις χώρες στις οποίες εφαρμόζεται. Και μάλιστα με αυτό που κάνουμε, μάλλον θα κάνουμε ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Πέντε δευτερόλεπτα οικονομία κάνετε. Πολύ ωραία, μου άρεσε αυτό ο ανταγωνισμό. Uh, Merci Madame la Présidente. Euh, rapidement, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Premièrement. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλά υπόθηκαν ε, κάτι που μου είναι ιδιαίτερα η κορίνα αποφάσισε, αλλά οι ε, συντάκτες του Pack ε, είναι εδώ, θέλαμε να κρατήσουμε την αυτή γραμμή. Δηλαδή. Και ποια ήταν η γραμμή, να βοηθήσουμε το Συμβούλιο να κάνει κάποιους ε, μικροϋπολογισμούς, δηλαδή να επανέλθουμε σε μηχανισμούς αντεστραμμένη αυξημένη πλειοψηφία. Αυτό δεν θα ήταν συνεπές τα όσο φάσαμε στο Pack. Δεύτερον, Συμφωνώ απόλυτα με την ιδέα ότι θα πρέπει να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος αποφάσεων που είναι εξίσου θεμελιώδης με αυτές που αφορούν στην επιβολή ενισχυμένη εποπτεία και λοιπά πρόβλημα δεν είναι μόνο η Κομισιόν και το Συμβούλιο, αλλά είναι η παρέμβαση του Κοινοβουλίου. Αυτό το λέω επειδή είμαι βουλευτή, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Είμαι υπέρ μια ισχυρή επιτροπή ε, με με θάρρος, ε, θα παίρνει αποφάσει τι οποίε θα υποστηρίζει ενώπιόν μας κλπ. Πάνω σε αυτά τα θέματα θα πρέπει να παραμείνουμε συνεπεί. Δεύτερον, νομίζω πως η Ελίζα και ο Ζων Πολ αλληλοσυμπληρώνονται, διότι προτείνουν επιπλέον αυτά, από αυτά που πρέπει η Κομισιό το Ταμείο διάσωση και το κεφάλαιο 11. Διότι αν υιοθετήσουμε μέτρα του τύπου κεφάλαιο 11, δίχως να έχουμε κάνει τα πάντα για να βοηθήσουμε τη χώρα να ε, εξέλθει από την κατάσταση, μα αντιμετωπίζεται περίπτωση πάυσης πληρωμών ή χρεοκοπίας. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ώστε να παραμένει αυτό ως ίστατη λύση, ίστατη προσφυγή. Θεωρώ ότι οι δύο εκθέσεις αλληλοσυμπληρώνονται και θα πρέπει να κάνουμε τη σύνδεση μεταξύ αυτών, τουλάχιστον από πολιτική σκοπιάς. Ετοιμάζουμε τροπολογίες αλλά θα πρέπει να πούμε κάτι παραπάνω για το Redemption Fund και για τα ευρωομόλογα. Αυτό θα εξαταστεί στην πρώτη φάση του χάρτη πορεία και ευχαριστώ Λίτσα που το έθιξε. Και μια ερώτηση. Η ελληνική εμπειρία δεν θα έπρεπε να μα ε, βοηθήσει στο να προσθέσουμε στον μηχανισμό του κάπου μέσα στο κείμενο κάτι σχετικά με το πάγωμα των ε, ιδιωτικής περιουσίας στο εξωτερικό. Πραγματικά εκπλήσωμε που ζητάμε αλληλεγγύη στους Ευρωπαίους, αλλά δεν ζητάμε αλληλεγγύη στο εσωτερικό της χώρας. Δηλαδή, πιο πλούσιοι της χώρας πηγαίνουν και καταθέτουν τα χρήματά τους σε άλλες χώρες, είτε Ελβετία είτε αλλού. Πιστεύω ότι το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνεται άμεσα στην αρχή της διαδικασίας, θα ήταν χρήσιμο. Και ε, μια ερώτηση για την Ελίζα, διότι θεωρώ ότι από τη στήκη του Μάστριχτ και το πρωτόκολλο υπαρθμών 12 υπάρχει κάτι που δεν είναι σαφές για το ΑΔΑΗ. Μιλάμε για διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος. Συμφωνήσω ότι αυτό καλύπτει και την καταπολέμηση του ελλείμματος και του χρέους. Και διερωτώ αν θα μπορούσαμε μπορούμε να πάψουμε να χρησιμοποιούμε αυτό το, το, την ορολογία που είναι ένα είδος για να ασχοληθούμε με το πιο κατεπήγον, πιο σοβαρό που είναι το χρέος. Το μήνυμα λοιπόν θα ήθελα να είναι πιο ισχυρό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, να ξεκαθαρίσω ότι οι άλλοι ομιλητές έχουν τρία λεπτά, οι σκιώδεις είχαν τέσσερα λεπτά. Ε, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, να εκφράσω τις επιφυλάξεις μου σχετικά με τα προτινόμενα που την έκθεση Γκοζέσα. Το Κοινοβούλιο ψήφισε ένα ψήφισμα το οποίο καταδεικνύει ότι το περιεχόμενο της συνθήκης της 1ης Μαρτίου ήταν ε, άχρηστη περιττή σχέση με τις αποφάσεις που λάβαμε για το Six Pack. Και εδώ μας προτείνεται να μεταφέρουμε στο παράγωγο δίκαιο αυτό που απορρίψαμε σε εκείνο το ψήφισμα. Αυτή είναι μια πρώτη φύλαξη που θα ήθελα να εκφράσω και θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο σημείο όπου πραγματικά παίζεται τον ε, πειραματιζόμενους μάγους 0,5%. Αυτός ο χρυσός κανόνας ε, δεν βρίσκεται στο six pack και αν σήμερα υπήρχε δημοψήφισμα στα κράτη-μέλη θα ήταν όχι σε αυτόν τον χρυσό κανόνα. Και εσείς θέλετε να τον ε, εισαγάγετε από το παράθυρο ενώ δεν τολμήσαμε να το συζητήσουμε στο πλαίσιο του Six Pack. Εξάλλου αυτό το θέμα το ανέφερε και σήμερα το πρωί, δεν έχω το χρόνο εδώ σήμερα. Τόσο κανόνα δεν έχει έννοια παρά μόνο εάν ε, μπορούμε να ανοιχνεύσουμε ένα διαθωτικό έλλειμμα το οποίο μακροχρόνια δεν αλλάζει και που ανταποκρίνεται στο το ποσοστό ανάπτυξη οικονομίας. Δεν έχει νόημα παρά μόνο εάν κάτι συμβαίνει. Και τότε το τρέχον έλλειμμα μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με την κοιμάση της συγκυρίας και μπορούμε να φτάσουμε στο 30%. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αναγνωρίζει ίδια αυτό το διαφορετικό έλλειμμα, το οποίο εξελίσσεται μέσω ε, ε, ε, βραχυπρόθεσμα και εξελίχθηκε ε, λόγω της υποβάθμισης της ε, ζήτησης ε, που συνδέεται με την κρίση. Και αν υπάρχει εξέλιξη σύμφωνα με το ποσοστό ανάπτυξης αλλά και της συγκυρία, εάν λοιπόν θέλετε να μειώσετε αυτό το συγκυριακό έλλειμμα κόβοντας όλα τα μέσα τα οποία μας επιτρέπουν να δράσουμε επί της ζήτησης, δεν θα κάνετε τίποτα άλλο από το να το επιδεινώνετε. Διότι μπορούμε να το διευθετήσουμε μόνο ε, στηρίζοντας την ανάπτυξη. Και αυτό, το six pack είναι αυτό το οποίο μας επιτρέπει να ε, προωθήσουμε την ανάπτυξη. Και για μία σειρά από λόγους ε, θεωρώ ότι είμαστε αυτή τη στιγμή, μάλλον αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα, είναι ότι ε, οπλίζουμε ένα όπλο οκτάσφαιρο κατά της ε, ανάπτυξης και παράγουν συναδέλφους να το εξετάσουμε με πολύ προσοχή διότι εδώ παίζουμε τους μαθητευόμενους μάγους ε, και σε πολιτικό και σε οικονομικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, μπράβο σας. Ε, καλύψατε ακριβώς τρία λεπτά υπερβάνως. Ευχαριστώ. Και στις δύο εκθέσεις ε, βλέπω ότι υπάρχει βούληση για περαιτέρω πρόοδο. Στην Ελίζα είδα την ε, λογική του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, την αναφορά ε, στο άρθρο 148, την κατάργηση της υποχρέωσης εγγραφής στα συντάγματα. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω είναι θετικά στοιχεία. Όπως και στην έκθεση Γκοζές για την για τους μακροοικονομικούς όρους ε, και προϋποθέσεις νομίζω ότι είναι θετικές προτάσεις, αλλά τρεις παρατηρήσεις ε, σχετικά με τις τρεις εκθέσεις. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούμε το άρθρο 136, άρα είναι μια ευκαιρία πολύ σημαντική για να επιλύσουμε το προβλήματα της ζώνης ευρώ. Το παίρνει λοιπόν ο διακύβευμα είναι αν με αυτό το διάβημα ανταποκρινόμαστε στι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ζώνη ευρώ. Και εγώ, μάλλον εμείς το είπαμε όταν συζήτησαμε το six pack, δέκα χρόνια ζώνη ευρώ μα έμαθαν ότι η μακρο, τα μακροοικονομικό δεν μπόρεσαν να ε, διορθωθούν ούτε με την, ούτε με την αναθεώρηση ούτε με καμία άλλη πράξη. Και με αυτόν τον τρόπο δεν ε, δίνουμε απάντηση και αυτό είναι το μόνο ερώτημα που θα πρέπει να μας απασχολεί διότι ακολουθήσουμε την Κομισιόν για να σε μια κατεύθυνση που δεν μας κάνει παρά να ανταποκρινόμεθα στην ε, προβλήματα της αγοράς αντί να αναρτηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα και τις επενδύσεις σε κάποιες στρατηγικές για την κατάργηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και ανισοτήτων. Και έτσι μπαίνουμε σε ένα νεφέλωμα νομικό το οποίο είναι αντιπαραγωγικό. Όλοι το ξέρουν, όλοι είμαστε απογοητευμένοι, απελπισμένοι. Κανείς δεν είναι σε θέση να μου πει ποιοι είναι οι κανόνες που, πώς εφαρμόζονται, με τι συνέπειες, πώς μια εθνική κυβέρνηση κυβερνά την ε, οικονομική του πολιτική με βάση αυτό τον ε, νομοθετικό πίνακα. Και από αυτή την άποψη λοιπόν ε, επανέρχομαι στα δύο ουσιαστικά ζητήματα. Πρώτον, όταν η διεθνής, το Διεθνές Σύμφωνο υπογράφηκε συμφωνήθηκε ότι η ανάπτυξη δεν περιλαμβάνεται και η Κομισιόν βγήκε με μια πρόταση από το καπέλο της. Ε, δεν θα έχουμε καμία συνέπεια ότι θα εξετάζουν τα δύο αυτά κείμενα. Και πολλοί συνάδελφοι μίλησαν για δημοκρατία και ανησύχησαν για το δημοκρατικό έλλειμμα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στη συμπερίληψη αυτών των δύο κειμένων. Αλλά το πρώτο δημοκρατικό έλλειμμα, δώστε μου ακόμα τρία το παρακαλώ. Το βασικό δημοκρατικό έλλειμμα είναι ότι ε, κυκλωθήκαμε από μία πρόταση κάποιων κρατών μελών για να συντάξουμε μία νέα συνθήκη τις οποίες δεν συζητήθαμε με το περιεχόμενο και τις εξελίξεις. του συνάδελφος Άγκροντ που να θεωρεί ότι τα στοιχεία αυτής της ε, συνθήκης δεν είναι οικονομικά βάσιμα και εμείς τι κάνουμε, τα συμπεριλαμβάνουμε στο παράγωγο νομοθεσία ενώ πρόκειται για συνθήκες που δεν έχουν ακόμα υπογραφεί και πόρο απέχουν από το να ακυρωθούν. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε αυτά τα δύο έγγραφα και να πούμε. Δεν είναι ο τρόπος για να, βγούμε, να βγει η ζώνη ευρώ από την κρίση. Ζητήστε από την Κομισιόν μια άλλη πρόταση που να βάνει υπόψη τα, τις μακροοικονομικές Αυτά. Ο Γκούναρ. Uh, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η δική μου προσέγγιση είναι κάπως διαφορετική από αυτήν των Γάλλων συναδέρφων. Πρέπει να πω ότι νιώθω ε, την γαλλική, το πνεύμα της Γαλλικής Επανάστασης ε, και μάλιστα πολύ έντονα. Γι' αυτό ίσως να διστάζω να μπω στη συζήτηση, αλλά Νομίζω ότι αν μπω στη συζήτηση θα είμαι με το μέρος του κυρίου Γκοζέ. Πολλές από τις προτάσεις στην έκθεση είναι σημαντικές και πιστεύω ότι πρέπει να τις δούμε από μια συγκεκριμένη πλευρά. Κάποιοι από τους συναδέρφους είπαν ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε ε, τις συνέπειες των ελλημάτων μόνο ε, σκεπτόμενοι θετικά λέγοντας ως πολιτική ότι δεν είναι σημαντικά τα ελλείμματα. Νομίζω ότι ε, ε, είναι ευθύνη μας να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε ε, με πολιτικές αποφάσεις το γεγονός ότι είναι, καταστροφικές, ότι είναι καταστροφικά τα ελλείμματα. Και θα διαφωνήσω με δύο από τους Γάλλους φίλους, οι, τα ελλείμματα δεν δημιουργούν πλούτο, υπονομεύουν τον πλούτο και τα υπερβολικά ελλείμματα δεν ε, ε, δίνουν ορμή στην οικονομία, ε, εμποδίζουν την οικονομία να αναπτυχθεί. Κοιτάξτε γύρω σας. Παντού στην Ευρώπη όπου έχουμε υπερβολικά ελλείμματα, έχουμε στασιμότητα, οικονομική στασιμότητα και αρνητική δυναμική και υπονόμευση του πλούτου. Σημαντικό είναι λοιπόν για να προστατεύσουμε την ευημερία. Ε, είναι, είναι καλό να έχουμε ε, χαμηλότερα επιτόχια και δυστυχώς έχουμε κάποια πειράματα προς την κατεύθυνση που ανέφερε ο συνάδελφος. Όταν συζητάμε τα προβλήματα της επικουρικότητας, ε, σημαντικό είναι στις δύο αυτές εκθέσεις ε, να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε κανόνες και πολιτικές. Πρέπει να έχουμε σταθερούς κανόνες ε, τον οποίων ε, την εφαρμογή να μπορούμε να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε. Αυτά θα πρέπει να τα συμφωνήσουμε μαζί. Δεν θα πρέπει όμως να επιτρέψουμε να υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις πάνω σε διαφορετικές πολιτικές. Ε, η κυρία Περέ ε, και ο κύριο Ονόκα αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό. Μπορείτε να έχετε οποιασδήποτε πολιτική θέλετε στη Γαλλία, αρκεί να έχουμε ε, κοινά συμφωνηθέντε κανόνε. Και ε, αυτά τα δύο νομοθετήματα ε, κάνουν ακριβώς τη διάκριση ανάμεσα στους κανόνες που πρέπει να δημιουργήσουμε και στις διαφορετικές πολιτικές. Μπορούμε να έχουμε όποια πολιτική θέλουμε, αρκεί να ακολουθούμε στους ίδιου κανόνες. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ξέρουν. θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τους συζητητές για το έργο που επιτέλεσαν. Θα ήθελα να κάνω κάποια πιο γενικά σχόλια για τις εκθέσεις αυτές στην αρχή και μετά σου να περάσω και πιο συγκεκριμένα σημεία. Καταρχήν, οποιαδήποτε ανάλυση γίνει θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γενικές ε, προϋποθέσεις ε, το ε, λεγόμενο six-pack, το δημοσιονομικό σύμφωνο και το γεγονός ότι καταβάλλεται σημαντικότερη εργασία τώρα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τη σχετική νομοθεσία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να πείσουμε τους πολίτες ότι δεν ε, ξανά και ξανά προτείνουμε τα ίδια πράγματα. Πρέπει επίση να εξασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία είναι συνεπής. Όλα αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα με το six-pack, καθώς επίσης και με ο... οποιασδήποτε άλλες ε, διακυβερνικές συμβάσεις. Ταυτόχρονα αυτή η λύση δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά πολύπλοκη ή διπλωματική. Εγώ είμαι ε, δικηγόρος, όπως και ο Ζοπόλ. Οι δικηγόροι λατρεύουν τους πολύπλοκους νόμους γιατί όλοι πρέπει να έρχονται να τους ζητάνε διευκρινήσεις. Εδώ πρέπει να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε κάποια δεσμικά όργανα, διαδικασίες κλπ. για τις οποίες θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς και αποτελεσματικές ε, λύσεις που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν κοινοβουλευτικά και δημοκρατικά στοιχεία, όπως τόνισαν και πολλοί από τους προελίσσοντες συναδέλφους. Εν κατακλείδη δηλαδή, αυτή η νομοθεσία θα πρέπει να είναι συμβατή με το six-pack, να είναι δημοκρατική και να είναι πρακτικά εφαρμόσιμη. Τώρα, συγκεκριμένε παρατηρήσει. Καταρχήν για την έκθεση Κοζέ. Υπάρχουν νομίζω εκεί κάποιε καινούριε θετικέ ιδέε. που δίνουν τη δυνατότητα νομικής προστασίας για τις διάφορες χώρες. Ίσως θα μπορούσαμε να, πραγμα... να εξετάσουμε περαιτέρω την ιδέα αυτή και επίσης να δούμε τι θα γίνει για τις χώρες ειδικές δυσκολίες σύμφωνα με το 7α. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι στο σώμα του κειμένου για να τα εξετάσουμε καλύτερα. Έκθεση κυρία Φερέρα τονίζει τη σημασία της ε, πρότασης ε, λύσης της Κομισιόν που μπορεί να ζητήσει από τις χώρες να ζητήσουν τη βοήθεια. Αυτό θα πρέπει να είναι επίσης κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να είναι δημόσια δηλαδή αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ όλους. Ο κάθε ένας από τους ηγητές μπορεί να πάρει τώρα τέσσερα λεπτά. Ξέρω ότι σε τέσσερα λεπτά δεν μπορείτε να τα απαντήσετε όλα, αλλά ίσως ορισμένα πολύ σύντομα σχόλια, από όλα. Ναι, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους εκείνους που εξέφρασαν παρατηρήσεις ή και κριτικές που είναι πάντα χρήσιμες. Δεν πρόκειται να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Μόνο λίγα. Για τον κύριο Χουντή, που συχνά διαφωνούμε, με ερώτηση ποια είναι η έννοια που δίνει στην τροπολογία 3. Μα η τροπολογία 3 έχει σαν στόχο να διαγράψει την ενδεχόμενη κύρωση για τα περιφερειακά ταμεία. Νομίζω ότι αυτό είναι σύμφωνα με αυτό που επιθυμείτε κι εσείς. Ερώτηση της Ιλβή. Όσον αφορά το πάγωμα των ε, ε αποθεμάτων ε, στο εξωτερικό. Υπήρχε νομίζω στο παρελθόν η δυνατότητα να παγώσουν στην Ευρώπη τα περιουσιακά στοιχεία κροτών που δεν ήταν πολύ, ε, πολύ συνεργάσιμα. Δεν καταφέραμε τίποτα. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Ιδίως αν πρόκειται και για χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί υπάρχουν τα ε, χρήματα. Αν σκεφτεί κανένα στην Ελλάδα, ε, τα προσωπικά αυτά στοιχεία βρίσκονται κυρίως στην Ελβετία και στη είπα. Ε, λοιπόν, το πρόβλημα είναι ακόμη πιο πολύπλοκο. Το θέμα της νομικής προστασίας. Είπα προηγουμένως ότι βασιζόμουν να ακούσω τις ιδέες των ΜΕΝ και των ΔΕ για να μπορέσω να διευκρινίσω και να οργανώσω τον δημοκρατικό έλεγχο της κατάστασης που ομολογώ είναι κάπως βία, που ανταποκρίνεται όμω σε κάποια ε, αναγκαιότητα που υπάρχει σήμερα και θα πρέπει να αναρωτηθούμε για την αποτελεσματικότητα τη ε, λειτουργίας και αντίδραση τη Ευρώπη προς την Ελλάδα. Γιατί εάν είμαι σωστά ενήμερο για την Τρόικα, ο εκπρόσωπος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τρόικα είναι τμήματάρχης. Δεν ξέρω τώρα ποιες είναι οι ικανότητες του ατόμου αυτού, κατά πόσο μπορεί να έχει με τις ε, ε, ε αρχές ε, και με την κυβέρνηση της εν λόγω χώρας τη συζήτηση στο σωστό επίπεδο. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να δημιουργηθεί πλούτος βασιζόμενος ε, στα, στα ελλείμματα διαβάζω προσεκτικά τα στοιχεία ε, όλων των οικονομολόγων. Εγώ ένα πτυχίο έχω, δεν ε, είμαι ειδήμονας, αλλά ξέρω ότι εκείνοι που δεν προέβλεψαν τίποτα ξέρουν ποια λύση θα βρεθεί τώρα. Και συγκρίνοντας τους μεν με τους δε, είναι το ίδιο. Γιατί ο καθένας ξεκινάει από αλλού και καταλήγουν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου που υπερψήφισα, σας το λέω, το ψήφισα. Αυτό το ψήφισμα έλεγε ότι εκτιμάται περιττό να περάσουμε από μία συνθήκη για να έχουμε στοιχεία οικονομικής διακυβέρνησης. Δεν είπαμε ποτέ νομίζω στο ψήφισμα αυτό ότι η ιδέα της οργανωμένης ε, ε, οικονομική διακυβέρνηση δεν ήταν καλή. Εγώ είπα μόνο ότι δεν χρειάζεται καν νέα συνθήκη. Ευχαριστώ και δεν ε, εκμεταλλεύτηκα τα τέσσερα λεφτά. Ευχαριστώ, ναι, δεκα ε, δευτερόλεπτα σου είχαν μείνει. Θα περάσουμε στην Ελίζα τώρα. Παρακαλώ, Ελίζα. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στη συζήτηση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία ή τέσσερα σημεία στο Ιγελ Πόρτας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να διακρίνουμε ε, τι είναι το δημοσιονομικό σχέδιο και τι ο δημοσιονομικός νόμος. Ε, υπάρχουν διάφορα στοιχεία στους προϋπολογισμούς. Ε, οι προπολογισμοί αυτοί όμως δεν μπορούν να λειτουργούν εκτός του ευρωπαϊκού νόμου. Το σχέδιο του προπολογισμού θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30 Απριλίου και μετά η Κομισιόν έχει χρόνο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Απ' την άλλη μεριά έχουμε τους ε, εθνικούς προπολογισμούς που βασίζονται στην εθνική νομοθεσία. Είναι σημαντικό αυτό που είπατε μεν, αλλά ε, θα πρέπει κάποια στιγμή αργότερα να το λάβουμε υπόψη μας. Ε, η ορολογία, ναι, η υπερβολικό έλλειμμα ε, χρησιμοποιείται εδώ σαν έκφραση. Και έχω την εντύπωση ότι είναι καλό να έχουμε αυτούς τους αυτόματους, ε, τα αυτόματα σημεία κίνησης. Η ιδέα του κυρίου Γκοζές να υπάρχουν όσο πάει και πιο πολύ αυστηροί κανόνες εποπτείας μιας χώρας όταν αυτή η χώρα συνεχίζει στην ίδια άγουσα και οδηγείται προς μια καταστροφή. Τώρα, η και κάποιοι άλλοι ερώτησαν κατά πόσον αυτό το κείμενο θα αντιμετωπίσει και θα λύσει τα προβλήματα. Όχι, προφανώς όχι. Ούτε το σεξπακ θα το κάνει αυτό. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, δηλαδή ή να απορρίψουμε τα πάντα, για παντός, ή από την άλλη μεριά να είμαστε πιο ο, ε, ανοιχτοί σε κάποιες τεχνικές λύσεις, να υπάρχουν κάποια ταμεία διάσωσης, να βρεθούν έτσι ε, λύσεις σιγά σιγά για τη διαδικασία ε, η οποία που εντάσσεται στο six pack παραδείγματο χάρη και στη μακροοικονομική ε, λύση. Να βρούμε μια λύση παραδείγματο χάρη για την έλλειψη αν θέλετε, συμμετρίας. Δεν θέλουμε να έχουμε διαφορετικές διαδικασίες εκάστοτε. Όλα αυτά θέλουμε να είναι ενωμένα, να υπάρχει μια συνοχή, γιατί αλλιώς οι κανόνες της δημοσιονομικής πειθαρχίας θα εφαρμόζονται ετήσια μεν, αλλά όχι μακροπρόθεσμα. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι να εξασφαλίσουμε να μην υπάρχει ριζοσπαστική απόκληση από τις δύο διαδικασίες. Υπάρχει βέβαια ένα πολιτικό θέμα, το 0,5% στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο, αν θα χρησιμοποιηθεί ή αν δεν θα χρησιμοποιηθεί. Αυτό όμως είναι κάτι που απαιτεί περαιτέρω συζήτηση. Χωρίς να είναι αυτό το κεντρικό σημείο της έκθεσης του κυρίου Γκοζές. Και αυτό που προτείνει νομίζω για το ε, κεφάλαιο 11, τον είπα, είναι σημαντικό. Από την άλλη μεριά όμως, ε, πρόεδρε, χρειαζόμαστε μια διαρθρωμένη προσέγγιση στην ε, ε, πρόταση Κομισιόν για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ε, να τις εξετάσουμε προσεκτικά και να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Να δούμε ποια είναι τα διδάγματα του παρελθόντος και πώς θα τα εκμετωρθούμε για το μέλλον. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που τηρήσετε και το χρόνο σας. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 5 Μαρτίου, στις 5 το απόγευμα. Όχι αργότερα, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε τις μεταφράσεις των κειμένων 11 για την εξέταση των τροπολογιών αυτών. 5 Μαρτίου λοιπόν. If we, we, could go to the 7th of March. Θα μπορούσαμε να, να πάμε μέχρι τις 7. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε στις 20 Μαρτίου να εξετάσουμε τις τροπολογίες και να ψηφίσουμε. 5 Μαρτίου ας πούμε τώρα και να δούμε αν μπορούμε να αλλάξουμε όλο το χρονοδιάγραμμα. Αυτή τη στιγμή πέντε. No, I know it's very short. Ξέρω, ξέρω δεν υπάρχει πολύ χρόνο. Είναι τρελά όλα αυτά στην Επιτροπή μας πάντα. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Εάν καταφέρουμε κάτι θα σας δώσουμε καινούρια ημερομηνία, αλλιώ πέντε.